So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's uh, go ahead with our intermeeting. Item 11 is a really important one. It is dealing with the G20 initiative for the Global Forum on Steel. Overcapacity. Μιλάμε τώρα για την υπερπαραγωγή του χάλιβος, λέει ο πρόεδρος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα είπαμε και την τελευταία συνεδριασή μας γιατί είχαμε την ε, συνάντηση κορυφής στο Buenos Aires Οπότε παρακαλώ τον συνάδελφο που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι έγινε στο Buenos Aires, στο G20. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η συνάντηση κορυφής αποτέλεσε την δέκατη επέτειο της πρώτης συνάντησης των G20. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχουμε όλο ένα και περισσότερες εντάσεις εμπορικές Έχουμε συγκρούσεις σε επενδύσεις και εμπόριο μεταξύ των πρωταγωνιστών. Δεν μπορέσαμε να έχουμε κάποιο είδου συνένεση στην Υπουργική Σύνοδο του Μαΐου και στο ΑΠΕΚ πρόσφατα. Οπότε η κοινή δήλωση τελικά ήταν μια επιτυχία για τους G20. Πάμε για έναν κοινό παρανομαστή στο εμπόριο και για πρώτη φορά δεσμεύτηκαν οι ηγέτες για μια μεταρρύθμιση του ΠΟΕ πιο εύρυθμη λειτουργία εν ώψη της επόμενης συνάντησης κορυφής. Αυτό ήταν προτεραιότητα και εμείς κάναμε διαμεσολαβητικές προσπάθειες έντονες. Οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με γίνοντο το κομμουνικέ, την ανακοίνωση ε, αφορούσαν την κόντρα Αμερικής Κίνας όσον αφορά τις ευθύνες για το σύστημα εμπορίου. Δεν ήταν δυνατόν να επαληθεύσουμε βέβαια τα παλαιότερα συμπεράσματα από το G7 και επίσης την δέσμευση να καταπολεμηθεί ο προστατευτισμός να είναι ανοιχτέ οι αγορές και να υπάρχουν δίκαιοι όροι. Ο πρόεδρος ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και μας παρέμβασε στις προτάσεις του Σεπτεμβρίου στον ΠΟΕ. Ήταν ένα θέμα διαφάνειας των σχετικών κοινοποιήσεων. Επίσης είχαμε παλαιότερες προσπάθειες της Μάλστρομ και του κυρίου Κατάινεν ούτως ώστε οι G20 να μειώσουν την παραγωγή του χάλιβα και επίσης να περικόψουν τις επιδόσεις που είναι η αιτία. Εξασφαλίσαμε σχετικές συστάσεις που συμφώνησαν οι Υπουργοί στο Global Forum για αυτή την περιπαραγωγή για πρώτη φορά εγκρίθηκαν από τους ηγέτες και τον Ιούνιο του 2019 θα γίνει μια έκθεση σχετικά με αυτό. Πάμε τώρα για την Ιαπωνική Προεδρία του G20. Γίνονται επαφές για την υλοποίηση της ε, διαγέρυξης του Buenos Aires. Γίνονται διεργασίες και στο G20 και στο Buenos Aires. Εδώ δίπλα έχω τον συνάδελφο Πέρεθ Κανιάδο που ήταν εκεί ε, και από τον Δεκέμβριο παρακολουθεί το τι γίνεται με αυτή την υπεραπαραγωγή του Χάλιβος να σας κάνει μια ενημέρωση, αλλά πρώτα πρώτα δύο λόγια όσον αφορά την ομάδα εργασίας του G20 που έγινε την περσμένη εβδομάδα στο Τόκιο. Εδώ η Προεδρία είχε φιλόδοξη μέσα σε διάταξη, όλα τα έγγραφα έχουν διαβαστεί στην Επιτροπή σας και το θεματολόγιο αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες του ΠΟΕ και όσον αφορά το σχετικό θεματολόγιο όσον αφορά τις τρευλώσεις στην αγορά είπαμε να θωρακίσουμε τους διεθνούς κανόνες και να συνεχιστούν οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο όμως στο Τόκιο φάνηκε ότι ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια οι περισσότεροι που ήταν υπέρ του θεματολογίου ε, θέλουν μία αναγκαία μεταρρύθμιση στον ΠΟΕ. Όμως κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση μόνο όσο χρειάζεται. Άρα να είναι η μικρότερη δυνατή μεταρρύθμιση. Άρα θα χρειαστεί να τους τα εξηγήσουμε τους επόμενους μήνες, θα χρειαστεί να πείσουμε κάποιους εκ των πρωταγωνιστών, να τους πούμε ότι πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση στον ΠΟΕ και ε, Εάν δεν γίνουν κάποιες βαθιές γενναίες αλλαγές στον ΠΟΕ, αυτός κινδυνεύει. Κινδυνεύει ίδια του η ύπαρξη. Τώρα να δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο τον Φρανθίσκο Κανιάδο για να σας ενημερώσει. Ευχαριστώ δύο λόγια για το Παγκόσμιο Φόρουμ σε ό,τι αφορά τις ε, ικανότητες πρόσβασης ε, να σας ε, κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή του 2016 και τότε λόγω της κρίσης που είμαστε τον κλάδο μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέρτωσε ένα σχέδιο αντιμετώπισης ε, της κατάστασης. Αυτό το συνολικό λοιπόν σχέδιο κάποιες πολιτικές, περιλάμβανε κάποιες πολιτικές, ε, εμπορικές, κάποια εργαλεία, κάποιες δραστηριότητες προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και για να αποφύγουμε αθέμητες πρακτικές, αλλά και σε αναγνώριση φυσικά του γεγονότος ότι αυτές οι δράσεις δεν πρόκειται να καταπολεμήσουν τις ε, βαθιές ρίζες της υπερπαραγωγής. Αυτό ήταν θέμα ε, διαφορετικών ε, κυβερνήσεων, κυρίως τη Κίνας, ε, που είχαν δημιουργήσει συνθήκες ε, υπερπαραγωγή. Αυτό πραγματικά διακύβευε την επιβίωση του κλάδου μας. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τις βαθύτερες αιτίε αυτές. Καταρχάς, ο πιο αποτελεσματικό τρόπος είναι οι πολυμερει παγκόσμιε προδιαγραφέ να καλύπτουν τι συνθήκε τη Κίνα. Προ το παρόν δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και εντωμεταξύ, εφόσον αυτό δεν γίνεται ακόμα, ήταν σημαντικό να υπάρχει ένα φόρουμ για να γίνεται μια συζήτηση, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τις πολιτικές. Φυσικά αυτό δεν είναι σκληρό εργαλείο, αλλά είναι πολύ ισχυρό παρόλα αυτά. Και αυτό γιατί αποτελεί τέκνο του G20. Ουσιαστικά λοιπόν ε, υποβάλλει αναφορά στην τελική ανάλυση στους ηγέτες του G20 και όπως ξέρετε για να πετύχουμε την προσοχή κάποιων συγκεκριμένων κυβερνήσεων όπως τη Κίνα και να πετύχουμε αλλαγή, χρειάζεται ε, η επιρροή της ε, κορυφαίας ηγεσία. Συγκεκριμένα τώρα, το Παγκόσμιο Φόρουμ το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη του 2016 έχει ουσιαστικά διάρκεια τριών ετών, έχει συμπληρώσει δύο έτη τώρα. Είναι χρήσιμο προς το παρόν για δύο λόγους. Καταρχάς, πετύχαμε ανεύ προηγουμένου επίπεδο διαφάνεια σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει στις μεγάλες χώρε παραγωγή ε, και κυρίως στην Κίνα. Ξέρετε ότι η Κίνα ήταν ε, μαύρο κυβότιο, black box, σε σχέση με το τι συνέβαινε σε ό,τι αφορά την παραγωγή, τι ε, ικανότητε παραγωγή. Τώρα υπάρχει μια βάση δεδομένων, η οποία τακτικά ενημερώνεται και τα δεδομένα για την παραγωγή, τι επενδύσει ανά σχέδιο στις 34 ε, χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Κίνας φυσικά. Τώρα λοιπόν πλέον μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Όταν η Κίνα κάνει υπόσχεση για τη μείωση της παραγωγής, αυτό φασικά είναι ε, πολύ κρίσιμο για την ε, καλή λειτουργία της αγοράς, κατά πόσο το κάνει ή όχι. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να επιλύθει το βασικό αυτό πρόβλημα το οποίο δυστυχώ επιμένει. Η διαφάνεια λοιπόν είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο μας βοήθησε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ε, κυβερνητικής μορφές ε, ενίσχυσης που αποτελούν πρόβλημα. Το φόρουμ λοιπόν αποτελεί μια χρήσιμη πλατφόρμα για ανοιχτέ συζητήσει και μια διαδικασία ελέγχου από ομοτήμους για οποιοδήποτε α, μέτρο που προκαλεί υπερπαραγωγή όχι μόνο στους κόλπους του ΠΟΕ. Αυτό προωθεί διάφορες, ε, μάλλον ε, ρίχνει φως σε διάφορες πρακτικές οι οποίες ως τώρα ήταν στο σκοτάδι, τις αγνοούσαμε και μας επιτρέπει, επιτρέπει στην διεθνή κοινότητα να ασκεί πίεση για σημαντικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επόμενα βήματα στα πλαίσια του φόρουμου. Φυσικά πρόκειται για το τελευταίο έτος. Μπορεί να υπάρχει παράταση. Θα γίνει μια συζήτηση για ενδεχόμενη παράταση. Στην επόμενη σύνοδο του G20. Αλλά ουσιαστικά δύο θέματα εξετάζουμε στα πλαίσια του φόρουμ. Καταρχάς, τη βελτίωση της διαφάνειας για κάποιες νέες μορφές ε, κρατικών ενισχύσεων που έχουν ανακύψει, κυρίως στην Κίνα να τις εξετάσουμε και να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στους ε, ομολόγους μας από την Κίνα για να κινηθούν προς την ε, πορεία της αγοράς και επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες ε, αναδυόμενες οικονομίες και άλλες επίσης εξελίξεις στις αγορές. Αυξάνονται λοιπόν οι διάφορες παραγωγές και καλό είναι λοιπόν να τα παρακολουθούμε όλα αυτά για να μην δημιουργηθεί εκ νέου μια κρίση υπερπαραγωγής. Αυτό θα είναι λοιπόν το σημείο εστίαση για φέτο. Αυτά λοιπόν συνοπτικά. Αυτά έχει ο κατάλογο, εκεί βρισκόμαστε. Και να σας πω ότι εδώ μας έχουν βοηθήσει πολλοί οι συνάδελφοι του ΩΣΑ, παρόλο που το φόρουμ δεν είναι φόρουμ ΩΣΑ, παρόλα αυτά λοιπόν μας έχουν βοηθήσει στις συζητήσεις, στην ανάλυση. Ήταν πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι ήταν και αυτοί μαζί μας. Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε ιδιαίτερος το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι συνεχιζόμενες αυτές ε, διαταραχές ε, και στρεβλώσεις της αγοράς να απειλούν τις ε, συνθήκες εργασίας μας και τον κλάδο μας ολόκληρο. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Αν σωστά κατάλαβα, έχετε πλέον όλα τα αριθμητικά στοιχεία για όλη την παραγωγή χάλιβα σε όλα τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τις εξελίξεις, τα στοιχεία, για παράδειγμα, τα δεδομένα στην Κίνα. Υπάρχει η φήμη ότι ε, μειώθηκε το, η παραγωγή χάλαβα το 2017 κατά 100 εκατομμύρια τόνους. Το 2018 30 έως 50 εκατομμύρια τόνους μείωση της παραγωγής. Τι λένε λοιπόν τα στατιστικά στα στοιχεία, για πείτε μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, η οποία θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό προκύπτει και από την ίδια την Κίνα, για την παρουσίαση των ε, αυτών, γιατί υπήρξε μείωση 50 εκατομμυρίων ε, τόνων. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτό δεν αρκεί έτσι κι αλλιώ. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη η μείωση. Θα δούμε κατά πόσο θα τηρήσουν τη δεσμευσή του, ωστόσο. Αυτό που μας ε, καταδεικνύουν τα αριθμητικά στοιχεία είναι ότι παρά τα σχόλια από κινέζικη πλευρά. ότι αυτό το ποσό των 150 εκατομμυρίων τόνων είχε ήδη επιτευχθεί ω μείωση στα πλαίσια τη αναδιάθρωση, Α, δεν έχει επιτευχθεί αυτό ακόμα. Είμαστε περίπου σε τάξη μείωση 100 εκα, έως 110 εκατομμύρια τόνοι. Επίσης, ε, το φόρουμ μας ε, επιτρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των όγκων αντικατάσταση της παραγωγής. Οι Κινέζοι το παρουσιάζουν ως μείωση, αλλά ουσιαστικά είναι αντικατάσταση της παραγωγής από παλιές ε, νέες εγκαταστάσεις. Υπήρξε λοιπόν μια μείωση γύρω στο 10%, αλλά ακόμα πολλά θα πρέπει να συνεχίσουν, να συνεχίσουν και πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν. Χάρη στο φόρουμ, λοιπόν παρακολουθούμε τι γίνεται. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε ποιήσεις στους Κινέζους ομολόγους. Ε, πιστεύουμε έτσι και αλλιώς ότι τα 150 εκατομμύρια τόν είναι πολύ σημαντική μείωση. Αλλά βάσει της δικής μας εμπειρίας, με την δική μας αναδιάρθρωση του τομέα του Χάλιβα, κυρίως στην δεκαετία του 70, του 80 και όλος ιδιαίτερος του 90, αυτή η μείωση δεν είναι καθόλου επαρκής για να επανελθεί μια ισορροπία στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη μείωση στην Κίνα για να πετύχουμε την ισορροπία και αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε από κοινού με τους εταίρους μας για να συνεχίσουμε να ασκούμε for that report. I was just struck in November, Bernd and I were part of the delegation to, of the intercommittee to the OECD, where we talked about the Global Steel Forum with the OECD colleagues responsible. And one of the comments which was made from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 Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μεταφέρουμε την επιθυμία αυτή στο υψηλό ε, επίπεδο λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. αλλά όπως είπε ακριβώς ε, το ε, μέλος του Κοινοβουλίου, κάθε Προεδρία στα πλαίσια των δυνατοτήτων τις οποίες έχει Αυτή θα αποφασίσει αν θα πραγματώσει ακριβώς την επιθυμία σας αυτή. Πάντως η συνάντηση στο ε, Buenos Aires ήταν μάλλον προτιμότερη, ήταν καλύτερη θα έλεγα από τις προηγούμενες και έγιναν, αν θέλετε, δόθηκαν κάποια μηνύματα τα οποία αντίστοιχα μηνύματα στο παρελθόν δεν ελαμβάνονται υπόψη. Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε μια συνολική λύση για τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Περνάμε στο σημείο 12 τώρα. Το σημείο 12 είναι η παρουσίαση του Υπουργού Εργασίας ε, της Ρουμανίας που προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών because of the uh, snow. I had also I had also delay in the morning, so <laughs> okay. it's quite common with the weather. So. Yeah. So. Ο πρόεδρος, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια σκληρή προεδρία γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος λόγω του πέρατος της ε, θητείας. Πάντως, έχουμε προκλήσεις σημαντικές να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και γονιούμε να μάθουμε τι θα κάνει η Ρωμανική Προεδρία. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω μερικά πράγματα που θα ήθελα να διαφωτιστώ, να με διαφωτίσετε. Υπάρχει ένα θέμα κορυφές προτεραιότητες για το κοινοβούλιο. Η, ο έλεγχος των εξαγωγών θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει γιατί είμαστε έτοιμοι. Προς το παρόν. Πάντως δεν έχουμε μπορέσει να πετύχουμε τον αναγκαίο συμβασμό. Ελπίζω να κάνει ό,τι μπορεί η Ρουμανική Προεδρία. Ούτως ώστε να αποκτήσει μια δημοτική θέση του το Συμβούλιο και να πάμε για κάποια συμφωνία πριν τις εκλογές. Τώρα, έχουμε επίσης τις εμπορικές συμφωνίε με Σιγκαπούρη και Βιετνάμ. Πέστε μα. που έχουμε φτάσει ω προ αυτό. επίση έχουμε και το θέμα των εμπορικών σχέσεων με τις ΕΕ γιατί την Παρασκευή είχαμε το σχέδιο της εντολής για τις επαφές, για τις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει η Προεδρία να εξασφαλίσει την ενότητα των ε, κρατών μελών. Για τον Brexit είναι γνωστές οι δύο επιλογές. Ίσως πρέπει να ετοιμάσουμε κάποια σχετική νομοθεσία, να γίνουν και εκεί κάποιες εμπορικές δημοκρατές, αλλά και εδώ θα πρέπει να ψηφιστεί, να αποφαστεί κάποια εντολή. Και βέβαια πάντα με διαφορετικέ διοργανωτικέ διαπραγματεύσει όσον αφορά εξωτερικέ πολιτικέ, όσον αφορά την κοινοποίηση των ενημερωτικών ε, γράφων. Άρα, πλούσιο το θεματολογία μας και έχετε τις σκητάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριος Οπρέα. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Με τη το ότι βρίσκομαι εδώ, μέσω των ε, αξιότιμων κυρίων βουλευτών, να σας πω τις εμπορικές μας προτεραιότητες, οπότε και να ξεκινήσω ε, με μια εξομολόγηση. Ξέρετε, ήμουν γερουσιαστής. Και από αυτή την ιδιότητα είχα έρθει πολλέ στο Κοινοβούλιο και είχα πάρα πολύ αξιόλογε επαφέ με του ευρωβουλευτέ, κυρίω όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σήμερα, επομένω, νιώθω ότι με τιμάτε. Ε, αλλά και εγώ είμαι περήφανο που έχουμε εδώ ω Υπουργό να σα παρουσιάσω τι θα γίνει με την Προεδρία και το εμπόριο. Οπότε μια που έχετε τους ε, εξαιρετικούς σας ε, διερμηνείς να σας ε, μιλήσω τουλάχιστον σήμερα και στην διάρκεια της Προεδρίας μας στη μητρική μου γλώσσα. Μιλόρ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που σας απευθύνω το λόγο. Να σας πω ποιες είναι οι της Προεδρίας μας όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η Ρουμανική Προεδρία Θέλει να υπάρχει συνοχή, να διατηρήσουμε προ τα προσπίσουμε τις κοινέ αξίες. Είναι θέμα ε, ευρωπαϊκής ενότητας, ούτως ώστε να γεφυρώσουμε τα χάσματα που υπάρχουν ε, από τόπο σε τόπο, ε, μέσα στην κοινωνία και επομένως θα πρέπει να έχουμε μια κοινή απόκριση στις προκλήσεις που υπάρχουν και σε επίπεδο του διεθνούς εμπορίου. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι μια ισχυρή ένωση να είμαστε ηγέτες για τον εξυγχρονισμό του πολυμερούς διεθνού συστήματο εμπορίου. Θα πρέπει επίση να θωρακίσουμε τα συμφέροντά μας σε αυτό το επίπεδο, αλλά και σε διμερές επίπεδο. Τώρα για το πολυμερές επίπεδο, το σύστημα το οποίο υπάρχει βλέπω κάποιου κανόνε αλλά τώρα εφίσταται αυτό το σύστημα κάποιες ε, πιέσει κάποιες πιέσεις που δεν είναι μόνο λόγω εμπορικών συμφέροντων. Έχετε την αμφιβόλο η όλη ύπαρξη του ΠΟΕ. Αλλά εμεί με μία φωνή έχουμε ζητήσει να γίνουν κάποιε μεταρρυθμίσει συστημικέ. Το ζητήσαμε και πρέπει να συνεχίσουμε να το ζητούμε. Γενικά οι προτεραιότητε τη Προεδρία μα έχουν ε, συγκροτηθεί γύρω από τέσσερι άξονε. Πρώτα-πρώτα, πώ θα αναβαθμίσουμε το ρόλο τη Ένωση ω παγκόσμιου παίκτη στη σκακέρα. Επίσης θέλουμε να υπάρχει σύγκληση, να υπάρξει ασφάλεια και να έχουμε μια ένωση κοινών αξιών. Μπορούμε να γίνουμε ισχυρότερο ε, παίκτη εάν συνεχίσουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο και πρωτοπόρο ρόλο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Ε, ε προωθούμε τον εξυγχρονισμό, αλλά αυτό ε, με την επιφύλαξη του να παραμείνει ο ΠΟΕ στον ρόλο το οποίο έχει τώρα με τους κανόνες ε, που έχει τώρα σε παγκόσμιο εμπορικό επίπεδο. Βέβαια, ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει ο κόσμος. Οπότε ο εξημενισμός του ΠΟΕ θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασικό εργαλείο για το εμπορικό σύστημα. Η Προεδρία μας θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ούτως ώστε να ξεπεράσουμε το σημερινό έξοδο όσον αφορά τους ε, ορισμός και διορισμός των μελών του δευτεροβάθμιου ε, δικαιοδοτικού οργάνου. Ε, και άλλοι το πρεσβεύουν αυτό στον ΠΟΕ και έχουν αρχίσει ήδη τον Δεκέμβριο στο Συμβούλιο οι συζητήσεις. Είναι θετικό αυτό και επίσης ε, θέλουμε να έχουμε τριμερείς επαφές με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Ήδη έχουμε κάποια αποτέλεσματα. Ε, ήδη υπάρχει θέληση για διαφάνεια, για βελτίωση της συμφωνίας του ΠΟΕ. Επίσης ο διάλογος με την Κίνα είναι διμερής και σημαντικός για τη λειτουργία του ΠΟΕ, για τις διαπραγματεύσεις σχετικά και εκεί ελπίζουμε να, έχουμε μετά το Νταβός και για το ηλεκτρονικό εμπόριο θετική εξέλιξη. Όλα αυτά σας δείχνουν ότι εμείς αντιμετωπίζουμε τις ε, προκλήσεις, έχουμε πλάνο και θέλουμε να μας ε, βοηθήσετε. Έχουμε το σχετικό σας ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου και και έχουμε επίσης ε, και το περσινό ψήφισμα του ΠΟΕ στη συνάντηση με τα κοινοβούλια. Οπότε να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να δούμε τι θα γίνει με την πρωτοβουλία για τις επενδύσεις. Ως Προεδρία, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει ένα πολυμερές πλαίσιο για τις επενδύσεις και να μιλάμε με μία φωνή ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα θεσμικά όργανα, όλα τα κράτη-μέλη. Ε, να επεξεργαστούμε όλους τους φακέλους που υπάρχουν νομοθετικούς και μη. Και έτσι όλα αυτά να τα κλείσουμε στο εξάμεινό μας τέλος πάντων πριν το τέλος της θητείας. Και σκέφτομαι επίση το οργανισμό για τη διπλή χρήση, διαπραγματεύσει με Μερκοσούρ, Κίνα, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Βιετνάμ. Και οπότε συνεχίζονται οι προσπάθειε στο Συμβούλιο για συμφωνίε ελευθερού εμπορίου, για την προστασία των επενδύσεων, για το Βιετνάμ. Είναι προτεραιότητα για μα και ελπίζουμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε να υπογραφούν αυτέ οι συμφωνίε και σε σχέση με την επόμενη Προεδρία. Πάντως θέλουμε να βοηθήσουμε ε, πώς η εμπορική πολιτική θα βοηθήσει να υπάρξει περισσότερη σταθερότητα στη γειτονιάζουσα περιφερειά μας και κυρίως προς ε, Ανατολά σε σχέση με την εταιρική σχέση. Το 19 θα είναι σημαντικό για αυτή την ε, περιοχή της Ευρώπης. Θα έχουμε και τη δέκατη επέτειο αυτής της πολιτικής εταιρική σχέση. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει περισσότερη πολιτική σύνδεση, ε, να βοηθήσουμε Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία και να υλοποιηθούν συμφωνίε ελευθερών εμπορίου να συμφίξουμε τις σχέσεις με Λευκορωσία και Αζερβαϊτζάν και Αρμενία. Επίσης και αυτό με την νότια γειτνίαση και να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία με την Τινησία ε, σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και αυτό είναι προτεραιότητα και είναι θετικό ότι η Κομισιόν ενέκρινε τις συστάσεις για, την διαπραγμα... τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την συμμόρφωση και άλλα εμπορικά θέματα οπότε η κοινή δήλωση είπα και Ένωση του Ιουλίου πέρυσι έγινε από Γιούνκερ και Τραμπ ε, ε, αυτή θα είναι η βάση για τις ε, επαφές. Πώ από αυτή την κοινή δήλωση τώρα θέλουμε να διαπραγματευτούμε για βιομηχανικά θέματα, για τους δασμούς, ε, τους δασμούς των βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης, η Ένωση θέλει να κάνει την πραγματεύση όσον αφορά το conformity assessment και όλα αυτά Επαναλαμβάνω, στη συνέχεια των πραγμάτων με τη ΣΥΠΑ. Στάνταρδελor și procedurilor τα Europene και Προσπαθούμε την τα πρότυπα, την διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα πρέπει όλα να γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Πρόκειται για έναν από τους στόχους της Προεδρίας μας. Να δούμε πώς θα καλύψουμε τους ε, πολίτες, όλους τους Ευρωπαίους έχουν προσδοκίες όσον αφορά το εμπόριο. Επίσης, θέλουν και διαφάνεια, αλλά βέβαια θα υπάρξουν και ωφέλης από την εμπορική πολιτική. Έχουμε μια σειρά από δημοσίες ε, διαβουλεύσεις. Αυτό να γίνει σε εθνικό επίπεδο, να γίνει με διαφάνεια. Με ΜΚΟ, διάφορους φορείς, ε, τις κυβερνήσεις. Βλέπετε ότι πρόσφατα μέσα από μια τέτοια διαδικασία ε, αναδείχθηκε ένας 15χρονος ως νικητής του σχετικού διαγωνισμού. Βλέπουμε επομένω πόσο οι αξίε ανδεικνύονται όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Άρα θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία ε, της κοινωνίας των πολιτών και των ε, Ευρωπαίων για τα θέματα της ε, χάραξης κοινής εμπορικής πολιτικής. Θα πρέπει το εμπόριο, θα πρέπει η εμπορική πολιτική να ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό σας το λέω ως υπουργό Εμπορίου, αλλά και ως υπουργό Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας στην κυβέρνησή μας. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι το 99% του συνόλου των ε, εταιριών στην Ένωση και δημιουργούν το 85% της απασχόλησης την τελευταία μας πενταετία. Και τα είπε πρόσφατα η Επίτροπος Μάλμστρομ. Οι ΜΜΕ δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα φόρα του διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει να ωφεληθούν περισσότερο οι ΜΜΕ αυτές. Αυτά θέλουμε. Και να τα έχουμε αυτά τα θέματα προτεραιότητα και να δούμε τι θα κάνουμε και με το Ρωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Να μην ξεχνούμε τα σημεία που σας είπα με βάση τις κοινέ αξίες της Ένωσης. Αυτά θα είναι το πνεύμα που θα διαπνέει την Προεδρία μας στο επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους ε, των πολιτικών ομάδων και μετά στα υπόλοιπα μέλη της ε, Επιτροπής. Νομίζω ότι τρία λεπτά μάξιμου μπορεί να έχει ο καθένα. Ο κύριο Φίσα από το ΕΛΚΑ. Θα μιλήσω ισπανικά, αν δεν σα πειράζει. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για την ξεκάθαρη και ευρύτατη ομιλία σας για το διεθνές εμπόριο, για όλα τα θέματα που θα χειριστεί η Προεδρία σας. Ε, δεν μπορώ να τα θίξω όλα, αλλά θέλω σε μερικά σημεία κάποιε διευκρινήσει. Πρώτα πρώτα, μα είπε για τι μεταρρύθμισει στον ΠΟΕ. Ναι, σημαντικό. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Τι γραμμή θα ακολουθήσετε για την μεταρρύθμιση αυτή. Έχετε πλάνο. Διαπραγματεύσουμε τη ΣΥΠΑ. Δυστυχώς για το TTIP τα πράγματα ήταν ένα ναυάγιο. Τώρα έχουμε τις επαφές της κυρίας Μάλμστρομ. Να δούμε πώς θα έχουμε διαπραγματεύσεις περιορισμένες στα βιομηχανικά, ρυθμιστικής υφής. Πώς το βλέπετε, τι περιμένετε, μια που έχετε λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να κλείσετε μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Επίσης, διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ. Ναι, όντως εκεί υπάρχουν προβλήματα. Α, και μετά αυτήν την συνάντησή μας θα συναντήσω κάποιους από την αθλητική βιομηχανία. Αυτοί ανησυχούν τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ. Είναι κάποια θέματα κοινωνικής πολιτικής γιατί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν τα πολιτερούν και πολλές χώρες. Τι λέτε, τι θα γίνουν αυτές τις διαπραγματεύσει. Εκεί μπορούμε να κλείσουμε τα θέματα σχετικά σύντομα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τώρα. Κύριε Σπινιερός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Καλή επιτυχία για την Προεδρία. θα ωφελήσει όλου. Θα είναι επιτυχία όλων. Και όλων για πέστε μα πιο συγκεκριμένα κάποια θέματα που αναδείξατε. Πρώτα πρώτα, πολύ βασικό. Διαπραγματεύσεις με τις ΙΠΑ. Σε τι πλαίσιο έγιναν διαπραγματεύσεις. Οι ΕΙΠΑ. έφυγαν από τα όσα συμφωνήθηκαν στο Παρίσι. Τι γίνεται με τα βιομηχανικά προϊόντα πολύ σημαντικό για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μεταρρύθμιση του πολιτού συστήματος για τη μεταρρύθμιση των κανόνων του ΠΟΕ. Εσείς τι θέση έχετε, τι γίνεται με το δεύτερο βάθμιο όργανο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αμεροληψία όσον αφορά τα μέλη αυτού του δικαστικού οργάνου. Τι γίνεται και... εδώ πέρα παίζονται συμφέροντα και τον είπα. Είπατε για εμπορικές συμφωνίες, είπατε ότι θέλετε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, μπράβο. Όμως, τα σχετικά κεφάλαια στις εμπορικές συμφωνίες έχουν κάποιες ρήτρες, δεσμευτικές, εκτελεστές. Τι θα γίνει, μπορούμε να βάλουμε κάποιες ρήτρες αναθεώρησης ούτως ώστε να θωρακίσουμε ε, αυτές τις απαιτήσεις για τε, τις ρήτρες που υπάρχουν, τις άλλες. Για την Λατινική Αμερική θα δώσετε προτεραιότητα στις σχέσεις μας. Λαμβάνομαι υπόψη. Όσον γίνονται σε κάποιες χώρες της κεντρικής Αφρικής, έχουμε, ε, συγγνώμη, Αμερικής. Έχουμε επίσης διαγωνιτεύσεις με το Mercosur. Θα το προχωρήσετε. Και έχουμε και το θέμα της καινούργιας και κατάστασης στην Βραζιλία. Για τη δική μας πολιτική ομάδα οι εξαγωγές διπλής χρήσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μπορούμε να αποσπάσουμε πριν τέλος της θετίας. Τέλος. Για την Αφρική θεωρώ ότι είναι στόχος προτεραιότητας. Θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα που είναι οι ρίζες, οι, οι αιτίες τέλο πάντων της μετανάστευσης. Τελικά το βιωτικό επίπεδο σπρώχνουν τους ανθρώπους να τρέχουν προς την Ευρώπη, να γκρεμίζονται από ένα τείχο ή να πνίγονται στη θάλασσα. Η κυρία θαλασσα κυρια από το ΕΣΥΑΡ. E ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπουργέ, και σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Είναι σημαντική αυτή η στιγμή και για μας, ε, γιατί θα έχουμε και τον Brexit, αλλά έχουμε και την Κίνα στον ΠΟΕ και ανησυχώ σε ό,τι αφορά την, ε, προτεραιότητε της ε, Προεδρίας. Πείτε μας λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της πολύ σημαντικής συνάντησης στη Γενέβη στον ΠΟΕ και επίσης οι διαπραγματεύσεις ε, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια. Σε ό,τι αφορά την Ασία τώρα, ελπίζουμε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιες συμφωνίες ε, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη να συμπεριληφθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα άλλες ε, συμφωνίες στην Ασία, θα δούμε οποιαδήποτε εξέλιξη υπό την Ορμανική Προεδρία όπως συμβαίνει συχνά, όποτε, όπως όταν μιλάμε σε τέτοιες συζητήσεις, όλοι έχουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να συζητήσω το θέμα της συμμαχίας ε, με την Αφρική. Πότε μπορούμε να αναμένουμε ότι θα προχωρήσει το θέμα αυτό, το προγραμματίζετε στην Προεδρία σας και φυσικά Σημαντικό είναι να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον των διαπραγματεύσεων και προφανώς και η Χιλή και το Μερκοσούρ αποτελούν σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ για τους ελεύθερους τώρα. Η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω τη Ρουμανική Προεδρία και τον Υπουργό Εμπορίου για την παρουσίασή του. Συγχαρητήρια και σας εύχομαι και κάθε επιτυχία σε ό,τι αφορά αυτές τις σημαντικές ε, εκθέσεις. Θα ήθελα να κοιτάξουμε και πιο ευραία ζητήματα ε, ανάπτυξη και την κατάσταση στην Αφρική. Αλλά είμαι βέβαιο ότι θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Να πούμε δύο λόγια σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ είναι πολύ συνεκτική και είναι σύγχρονη ω ε, συμφωνία, σύμβαση ελευθέρου εμπορίου και θεωρώ ότι θα βελτιώσει πραγματικά το εμπόριο μεταξύ των δύο περιοχών. Θα επιφέρει και κοινωνικέ εξέλιξει με θετικό τρόπο στο Βιετνάμ. Και αυτό γιατί υπάρχουν ε, κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης στη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να εγκριθεί στην θητεία αυτή η συμφωνία. Γιατί είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν σωστές ε, σχέσεις με το Βιετνάμ. Μόνο με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σε μια τεταμένη περιοχή στην Νοτιοανατολική ναι. Ασία, γιατί το Βιετνάμ θα έχει και πολλού ανταγωνιστέ στην περιοχή. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε την υποστήριξη της ε, συνθήκη αυτή. Ελπίζουμε να επιτευχθεί η συνθήκη αυτή το σύντομο δυνατόν. Ερωτώ λοιπόν, είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων σα, είναι στις πρώτε σα προτεραιότητε. Ε. Για την Γκουε τώρα ο Έλμουντ Σόλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον Υπουργό. Για την ε, καθιερωμένη αυτή παρουσίαση σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πολιτικές και τις πολιτικές επενδύσεων θα με ενδιαφέρεται από πλευρά μου να ακούσω το εξή, γιατί προφανώ είναι σημαντική η συμφωνία με το Βιετνάμ, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω είναι τι θα γίνει με τι υποχρεώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, και το περιβάλλον και την απασχόληση. Πώ θα λεφθούν όλα αυτά υπόψη, γιατί πιστεύω ότι η διαδικασία επικύρωση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πετύχουμε σημαντική βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης σίγουρα θα γνωρίζετε και τις καταγγελίες των ε, ΜΚΙΟ και από τα κρατημέλη αλλά και από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά δεύτερον, η Ρουμανική Προεδρία. Πώς θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση των πολυμερών ε, προδιαγραφών σε θέματα ε, εμπορίου, γιατί εδώ έχουμε σημειώσει τέλμα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια φρέσκια προσφέγγιση που ακριβώς ε, θα μπορέσει να προωθήσει την πολυμερία και το θέμα του σώματος αυτού τους κόλπους του ΠΟΕ και θα ξέρετε ότι και από πλευράς Κοινοβουλίου τίθεται το θέμα της μεγαλύτερης ε, συμπερίληψη των κοινοβουλίων της περιοχή. Αυτό θα ήταν το ευκταίο. Θα μπορούσαμε. μήπω η Προεδρία να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική ε, φάση και εμείς δεν θα είμαστε σε θέση όλες αυτές οι προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα να τι ελέγξουμε. Αλλά το νέο κοινοβούλιο φυσικά και θα κάνει τον απολογισμό. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει αμα, αξιοπιστία. Γιατί η αξιοπιστία είναι αυτή που μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προφανώς και για τις ευρωεκλογέ. Τέλος. Μία ερώτηση η οποία με απασχολεί και με το Βιετνάμ αλλά και με την Κίνα. Τι θα γίνει με την ε, Κίνα λοιπόν το θέμα των ε, κρατικών, ε, των δημόσιων ε, εταιριών. Υπάρχει μια έκθεση χώρας για την Κίνα, αλλά είχαμε ανακοινώσει ότι δεν είναι προκειμένο να καταστεί δίκαιο της Κίνας. Οτιδήποτε θέμα και των κρατικών επιχειρήσεων. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για το Βιετνάμ. Μήπως αναπτύσσουμε διπλά δύο μέτρα και σταθμά ή έχουμε κοινά πρότυπα. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει εδώ η Ρουμανική Προεδρία. Ο κύριος Σάλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι μόνιμος εισηγητής για την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ, στην οποία έγινε αναφορά επανειλημμένα. Η Ρουμανική Προεδρία έχει προτείνει τη συζήτηση για το θέμα αυτό στη συνάντηση ε, του Συμβουλίου τον μήνα Μάιο. Είναι σαφές ότι αυτό θα εμποδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή γιατί η τελευταία μας ολομέλεια είναι τον Απρίλιο. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα καθυστερήσει η απόφαση τουλάχιστον για ένα χρόνο. Έχουμε εκλογές, ε, μετά θα έχουμε ε, την ε, δημιουργία των μηχανισμών του νέου κοινοβουλίου και συνεπώς θα καθυστερήσουμε και θα πάμε για τον Οκτώβριο ουσιαστικά, κάτι το οποίο θα είναι αδικαιολόγητο. έστειλε επιστολή και σε εσά και στον πρόεδρο του στο Συμβούλιο ζητώντα την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να επιταχύνετε κάπως τα πράγματα, να επανεξετάσετε το χρονοδιάγραμμα και δεν θα πρέπει εμείς ε, να αφήσουμε να μας ξεφύγει χρονικά η διαδικασία αυτή εκεί των Darling. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μία ερώτηση η οποία τίθεται επανειλημμένα σχετικά με την εμπορική συμφωνία, την εταιρική σχέση με το Βιετνάμ θα καθυστερήσει, δεν ξέρουμε για πόσο θα καθυστερήσει Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να μας ε, ε, διαβεβαιώσετε ότι θα συμπεριληφθούν στη συζήτηση θέματα όπως τα εργασιακά δικαιώματα στο Βιετνάμ. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε κάποιες ε, νέες εξελίξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις στον Ταβός. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις σύντομα. Ε, θα δούμε τι θα γίνει και με τις διαπραγματεύσεις ΤΙΣΑ ε, που έχουν ε, προς το παρόν παγώσει. Θέματα τα οποία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν προκαλέσει πάρα πολλές δυσκολίες. Διερωτώμεθα λοιπόν αν πράγματι θα υπάρξει μια κάποια αλλαγή στις θέσεις σας. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέα που είναι μαζί μας σήμερα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όλοι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο Βιετνάμ. Όπως ξέρετε ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για μας. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε ε, στην ε, εταιρική σχέση με το Βιετνάμ το ταχύτερο δυνατόν. Μας ανησυχεί το ότι θα συζητήσετε το θέμα αυτό στις 28 Μαΐου. Διερωτώ με αν θα μπορούσατε να κάνετε τη συζήτηση αυτή νωρίτερα. Δεν ξέρω ποια προβλήματα είναι αυτά τα οποία σας εμποδίζουν να το κάνετε, αλλά καλό θα ήταν η συζήτηση να γίνει πραγματικά νωρίτερα. Το Κοινοβούλιο έχω την αίσθηση ότι όταν εξετάζει τα θέματα αυτά το κάνει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και σε μεγαλύτερο βάθος από ότι το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις τις οποίες μου θέσατε, λέει ο κύριος Σόπρεα. Είναι φυσιολογικό που θέτεται ορισμένα από τα θέματα τα οποία επανέρχονται στις διαδοχικές προεδρίες. Η Ρουμανική Προεδρία θέλει να είναι ε, φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική. Το θέμα δεν είναι ε, για τον Brexit η συζήτηση, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την 29η Μαρτίου αλλά δυστυχώς η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα γενικότερα στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω αν πάρουν οι πολίτες στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνω, τις απαντήσεις τις οποίες θα επιθυμούσαν. Ταυτόχρονα τον Μάιο έχουμε και τις ευρωεκλογές. Οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι σχετικά περιορισμένες και αυτό εξηγείται στο ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες οι προεκλογικές. Σε συνεργασία λοιπόν και με τον κύριο Λάγκερ και με τον κύριο Βίνκλερ στο, στο Ορμανικό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε καλά ποια είναι τα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις ε, δυσκολίες, τα προβλήματα. Και να ευχαριστήσω εδώ και την Αυστριακή Προεδρία για τον τριγωνικό διάλογο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες τις οποίες έκαναν έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτό συζητιέται αυτή αυτές τις μέρες στο Κοινοβούλιο όπως είπατε. Και ένα από τα θέματα ε, που είναι πολύ σημαντικό είναι ο μηχανισμός ελέγχου της συμφωνίας ε, και ε, οι συνέπειες των επενδύσεων Θα ήθελα λοιπόν να δώσω κάποιες ε, απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Στον Ταβός ε, τα θέματα αυτά είναι υποσυζήτηση. Ε, και θα γίνουν και κάποιες ανεπίσημες συναντήσεις στις, 32, στις 23 ε, και 24 ε, Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι. Η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε, κάτι το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιδιώκουμε την ενότητα δράσης. Προσπαθούμε να είμαστε ο ειλικρινής ενδιάμεσος, σε μπάση περιπτώσει, που θα βοηθήσει την επίτευξη του συμβιβασμού. Δεν θα εκφράσω λοιπόν ως Προεδρία τις ιδέες της που έχουμε σαν κυβέρνηση, αλλά ε, τις θέσεις των συναδέλφων που θα μπορούσαν ε, να, χρησιμοποιηθούν ως απαντήσεις στα ερωτηματικά τα οποία εσείς θέτετε. Νομίζω λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή που έχει ξεκινήσει θα πρέπει να συνεχιστεί, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και στα πλαίσια των τριμερών επαφών Ιαπωνίας, ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συναντήσεις αυτές υπήρξαν κάποια μικρά βήματα και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θεωρούνται απαραίτητα και από τις δύο πλευρές για τη σωστή λειτουργία των εμπορικών συμφωνιών. Έχω προσκαλέσει επίσης τις συναντήσεις μας και τον Γενικό Διευθυντή Αζεβέδο Υπήρξαν αρκετές πιέσεις σχετικά με το Βιετνάμ. Είναι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας και τα πράγματα θα πρέπει να εξελιχθούν σταδιακά. Ξέρετε πού βρισκόμαστε σήμερα και επαναλαμβάνω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ και γι' αυτό Περιμένουμε από το Βιετνάμ να επικυρώσει τα τρία πρωτόκολλα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Υπήρξαν επίσης και ε, προσπάθειες για την διαμόρφωση μιας νέας εντολής για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όπως είπα πριν, θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να κινηθούν ταχύτερα. Για να προχωρήσουμε με ταχύτητα όμως απαιτείται πνεύμα συνένεσης στα πλαίσια της συνάντησης του τέλους Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις με πολύ μεγάλη προσοχή. Επιμένουμε ότι η σημασία έχει η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφάνεια βέβαια. Και επαναλαμβάνω ότι τα θέματα της γεωργίας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση στην παρούσα φάση. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά. Θυμάστε πρόεδρε Λάγκε και τις συζητήσεις στο Βουκουρέστι. Έχουμε το θέμα της διπλής χρήσης, των προϊόντων διπλής χρήσης. Εδώ έχουμε κάποιες διαφορές. Σε ορισμένες χώρες τα θέματα αυτά ανήκουν στην αυμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου, ενώ σε άλλες στην αυμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως προσπαθούμε να συντονίσουμε το Συμβούλιο και να προκαλέσουμε μία έγκαιρα, να προκαλέσουμε μία συζήτηση στο Συμβούλιο. Τώρα για την Αφρική Γενικά έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις. Ε, γνωρίζετε ότι σε κάποια σημεία υπάρχει συμφωνία. Πάντως τον Φεβρουάριο θα πάω στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος για ένα χρόνο θα προεδρεύει του οργανισμού ε, των Αφροκανικών χωρών και θα προσπαθήσουμε μαζί τους ε, να εντοπίσουμε τις θέσεις ε, τις δικές μας απέναντι στα θέματα που τίθενται ε, για την Αφρικανική Ήπειρο. Τώρα με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία τα θέματα αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος ε, ταχύτατα. Oh. <clears throat> Uh, uh, uh, Η κυρία Ροντρίγκε επίση ρώτησε για τη Μερκοσούρ. Είχα μια συνάντηση χθε ε, το πρωί με τον ε, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Μερκοσούρ ε, και συζητήσαμε τα θέματα αυτά. Προσπαθήσαμε να αποκρισταλώσουμε τι απόψει μα. Είχαμε πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία. Στη φάση αυτή τώρα όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε Ποιε είναι οι απόψει των άλλων πλευρών. Ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε καλή πρόοδο και στα θέματα Μερκοσούρη. Σίγουρα είναι στην ατζέντα μας αυτό το θέμα. Uh, uh, και επίσης ακούσαμε μια ερώτηση για τις... Ε, Thank you. Της κυρίας ε, Και όντως θα είναι ένα από τα θέματα που ελπίζουμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και εδώ θα θέλουμε να διευκρινίσουμε το θέμα αυτό θα τεθεί και στη Γενέβη, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι κάθε μικροεπιχείρηση σήμερα μπορεί να είναι πολυεθνική, να εξάγει σε διάφορες αγορές από απόσταση. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα θέματα αυτά και να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ε, η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να έχουν ε, αρνητικέ επιπτώσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν τα είχαμε συζητήσει αυτά πριν από κάποια χρόνια. Πού να τα φανταζόμασταν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα σήμερα πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα φαντάζεται μπορεί να έχουν σημασία για τις νέες νεοφύσεις επιχειρήσεις ε, τα επόμενα χρόνια. Αλλά εκ παραλλήλου θα πρέπει να φροντίσουμε τι σημαντικές ε, αξίες που έχουμε ως Ευρωπαίοι. Αυτές λοιπόν αποτελούν και την, τις κατευθυντηρίες γραμμές για την Προεδρή μας. Αυτές οι κατευθυντηρίες γραμμές, αυτές οι αξίες λοιπόν. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τις γραμμές αυτές προς τη Γενέβη. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό Ανέφερα λίγο πολύ όλα τα ζητήματα. Okay. Thanks Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό. Περαιτέρω ερωτήσεις, αν όχι, να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ και υπολογίζω στην υποστήριξή σας, ε, λέει ο Υπουργό, και πραγματικά εκτιμώ το γεγονό ότι αυτές θέσατε ερωτήσεις και ελπίζω να ξαναβρεθώ στην Επιτροπή σας. Κύριε Λάγκε, όποτε επιθυμείτε και θα έρθουμε στην Επιτροπή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Okay. Point 13. Σημείο 13, λέει ο Πρόεδρος. Έκθεση για την ε, αντιπρόσωπια ad hoc στον ΠΟΕ στη Γενέβη. 6 και 7 Δεκεμβρίου. Έχουμε πάνω από 300 ε, συμμετέχοντες ε, από πολλές χώρες που πήραμε μέρος την ε, συνέλευση του ΠΟΕ, στη σύνοδο του ΠΟΕ. Η διάσκεψη οργανώθηκε από την Διακοινοβουλευτική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε την ε, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ναμίμπια, την κυρία Βιλίους και εμένα ως ε, συμπροεδρεύονται. Ο κύριος Καστάλτο έκανε μια ομιλία και ο κύριος Σταγιάννη. Και ύστερα έγιναν κάποιε πραγματικά καρποφόρες συζητήσει με τους εκπροσώπου του ΠΟΕ. Είχαμε και τον αντιπρόεδρο του ΠΟΕ και πολλούς άλλους προεξέχοντας. Στην φάση προπαρασκευαστική κάναμε και κάποιες εργασίες στην ε, καθοδηγητική επιτροπή. Ετοιμάσαμε ένα έγγραφο το οποίο και εγκρίθηκε. Διοργανωθήκαν κάποια πάνελ από τον κύριο Ριμπίχ και τον κύριο Σόλτς. Και κλείνοντας προέκυψε και ένα έγγραφο πορισμάτων. Συνολικά, θεωρώ ότι ήταν πραγματικά πολύ ζωντανή αυτή η εκδήλωση. Και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει πραγματικά εδώ πέρα σημαντικό ρόλο. Άλλα σχόλια τώρα από αυτού. Είμαι. Πάρα πολύ καλά. Άρεστα τα είπε ο πρόεδρος. Συμφωνώ με όσα μας εξήγησε και ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαγενοβουλευτική συνάντηση του ΠΟΕ και σε όλα τα φόρα που την συνόδευαν. Υπήρξε αυτή η τελική δήλωση, ε, υπήρξε ομοφωνία, φυσικά και έχουμε 164 χώρες με διαφορετικές ε, θέσεις, οπότε δεν είναι και λίγο αυτό που καταφέραμε. Μια συμφωνία που βέβαια δεν μας καλύπτει 100% αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα. Βήμα σημαντικό. Οπότε νιώθουμε ικανοποίηση σε σχέση με τη συμμετοχή μας εκεί βοήθησε πάρα πολύ η, η γραμματεία και νομίζω ότι με τις κοινέ προσπάθειες κάνουμε βήματα προόδου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχει άλλος παρατηρήσεις. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για το υπαριθμό 14. Το πρωί τα είπαμε. Σχέσεις με τις είπα; Εμπορικές σχέσεις. και εξηγήθηκε τι στρατηγική υπάρχει και σε σχέση και με την διαπραγματευτική εντολή της Παρασκευής. Ε, βέβαια και παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε ακόμα λεπτομερέστερα ποιες θα είναι οι συνέπειες της παρούσης πολιτικής τις σχέσεις τις εμπορικές ΕΕ αλλά και τις συνέπειες για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Οπότε για ακριβώς αυτό τον λόγο εκπονήθηκε μία μελέτη την συνέταξη ο κύριος Πίτερ Τσέις Νομίζω ότι μπορεί να μας ε, δώσει μια υποστημονική τεκμηρίωση για το θέμα αυτό. Κύριε Τσέις, έχετε το λόγο για την μελέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία Κάναμε με του συνεργάτε μου τη μελέτη αυτή. Ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, ξέρω ότι πιέζεστε γιατί έχετε πάρα πολλά θέματα αλλά και το πρωί με τον Γενικό Διευθυντή είχατε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Ήθελα κάποιε διαφάνειε λάβουν τα μέλη τη Επιτροπή, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Ήταν ε, για την μελέτη. Οπότε παρακαλώ δώστε του ε, αυτή την ε, παρουσίαση αργότερα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι γίνεται, τι έχει επιτευχθεί και επίσης προσπαθούμε να δούμε τι συνέπειε θα υπάρχουν για το υπερατλαντικό εμπόριο, τι γίνεται με το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου, να δούμε διαφορετικά σενάρια και σύντομα να προσπαθήσω όχι να ε, συζητήσουμε το τι έχει γίνει γιατί νομίζω ότι αυτά τα ξέρετε αλλά ήθελα να μιλήσουμε για το πνεύμα που διαπνέει την ε, κυβέρνηση των ΙΠΑ και να δούμε και τι σενάρια υπάρχουν και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Τώρα, για να δούμε. Τι ελαττήρια έχει για αυτή την πολιτική, είπα. Θεωρούν ότι είναι θύμα της εμπορικής συμφωνίας των εμπορικών σχέσεων και όχι ως θύμα ε, των προηγουμένων κυβερνήσεων. Αυτό που πιστεύουν είναι ότι για την βασική τους πολιτική, την προηγούμενη πολιτική τους θεωρούν ότι ε, ε, άνοιξαν την ε, πολιτική για να έχουν γεωπολιτικό πλεονέκτημα οπότε αυτό έγινε. Άνοιξε η αγορά τον είπα, αυτό πιστεύουν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ακριβώς για να υπάρχει να έχουν το πάνω χέρι γεωπολιτικά. Όμως η παρούσα κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει αυτή την πολιτική και έτσι τελικά έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική πολιτική για τις διαπραγματεύσεις οπότε ξεκινάνε λέγοντας τι θα, σας, τι θα μας δώσετε για να σας δώσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το πνεύμα όλων των διαπραγματεύσεων ε, αυτής της ε, κυβέρνησης και αυτό επίσης καταδεικνύεται από το εμπορικό έλλειμμα όπως δείχνει η διαφάνεια που σας διέβασα. Η Κίνα έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα για εμπορεύματα και για υπηρεσίες. Αλλά έχουμε 150 δις ε, τα οποία τα προκαλεί η, ε, το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ένα σωρό στοιχεία σε αυτή την ε, μελέτη, τι έχει γίνει, δεν θα το επαναλάβω. Αλλά να δούμε σήμερα που βρισκόμαστε, τι γίνεται σχετικά με τον ΠΟΕ και με την Κίνα. Ο κ. Τεμαρτή σας τα είπε, κατά το πρωί. Αλλά Σίγουρα οι δεσμοί για τον ε, Χάλιβα αυτό κάτι ήταν. Αλλά τελικά αυτό που κάνανε ήταν κάτι που χτύπησε τους ίδιους. Μπούμεραν για την Αμερική. Σας παραμείνω στις ε, παλαιότερες δηλώσεις τους και τον Οκτώβριο κλείσαμε τη μελέτη, αλλά από τότε έχουμε κάποια πρόοδο. Θέλουν να διαπραγματευτούν έθεσαν κάποιους ε, στόχους και η Επιτροπή ε, διερευνά τώρα το πώς θα βγει η δημοτευτική εντολή. Τα είπατε το πρωί ότι έχουμε δυόμιση χρόνια ε, για το TTIP που τα λέμε και τα διαμορφευόμαστε αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει χάσμα απόψεων θέλουν ευρύτερες ρυθμίσεις οι Αμερικανοί από τους Ευρωπαίους. Η Κομισιόν θέλει να επικεντρωθούμε στο conformity assessment και ε, στους δασμούς. Βέβαια ένα άλλο σημείο κλειδί και ακαθόδες είναι η γεωργία. Άρα να πούμε ότι στους στόχους τους που συνοψίζονται στις διαφάνειες που σας έστειλα έχουν και τις δημόσιες συμβάσεις Επίσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, για περιβάλλον, για απασχόληση και μας ζητάνε να είμαστε πιο αποφασιστικοί σχετικά. Όμως, τίποτα για το ISDS. Θέλουν άλλη ρυθμίση σε σχέση με τις διαμοντεύσεις του TTIP βασικό. Είπαν ότι θέλουν να γίνουν βαθμιά οι διαπραγματεύσεις για να υπάρχουν και διαβουλεύσεις με το Κογκρέσο. Πού πάμε, να δούμε τι σενάρια υπάρχουν. Βέβαια, το βασικό θέμα είναι, ε, βέβαια έχουν και αυτή την μελέτη ε, την αυτοβιομηχανία και το εθνικό συμφέρον. Δεν ξέρω αν θα δημοσιοποιηθεί και πότε. Α, το Φεβρουάριο. Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι θέμα εθνική ασφαλεία το ότι θα με την αυτοκινητομηχανία λένε ναι, και επίση να δούμε τι επιλογέ έχει ο πρόεδρο και τι θα κάνει με τι επιλογέ που έχει. Διότι λέγεται ότι μία από τι επιλογέ είναι να βάλουν στα ανταλλακτικά δασμούς, να προστατευτούν. Αλλά θα μπορούν να στοχεύσουν την υψηλή τεχνολογία, τα αυτόματα, αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο βέβαια είναι θέμα για τον Κινέζων. Εάν αυτό κάνουμε τους δασμούς, κυρία Μάλστον, κύριος Ντεμάρτη, ήταν σε αυτό κατηγορηματική, ότι η Κομισιόν επίσης θα είναι αδαμάντη, δεν θα ε, συνεχίσει τις ε, επαφές. Τα είπε ο κ. Δημοκρατία και μίλησε για αυτά τα 100 εκατομμύρια ε, προϊόντων των οποίων είναι βασικός προμηθευτής η Αμερική. Οπότε πάμε τώρα για 80 δις που θα πρέπει να ρυθμιστούν γιατί θα αφορά ματαιώσεις ε, μπορείς αυτοκινητών άλλα 10 ε, δις για χάρη. Τι θα γίνει, όλοι θα βγουν χαμένοι. μπορεί κανείς να έχει σταθερή θέση. Τι αντίπεινα θα λάβει ο Τραμπ. Βλέπετε, ε, έτσι έχουν οι δυναμικές κατάστασεις, ε, οπότε δεν θα πρέπει να κάνουμε να το πιστόλι στον κρόταφο. Θα πούμε ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας αλλά θα έχουμε σταθερή θέση και στις διαπραγματεύσεις υπάρχει κάτι λάθος το να επικεντρωνόμαστε στην γεωργία θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα άλλο η πρόσβαση στην αγορά και άλλο τα ρυθμιστικά και για τη γεωργία και πάρα πολλοί Ξεχνώ ότι είμαστε μεγαλύτερο εξαγωγέ. Είμαστε πάρα πολύ ισχυροί. Έχουμε τρομερό εμπορικό πλεόνασμα για τη Γεωργία όσον αφορά τη ΣΥΠΑ και για την πρόσβαση στην Αμερική. Για την πρόσβαση στην αγορά μπορούμε να τους κοντράρουμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουν ελεύθερη αδασμολόγητη πρόσβαση στην Γεωργία. Το θέμα πάντως δεν είναι ε, η ρύθμιση. Το θέμα είναι το SPS. Οπότε δεν θα πρέπει έτσι να ανατινάξουμε τους στόχους μας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, τα θέματα της διατροφικής ασφάλειας και τώρα τα ρυθμιστικά είναι άλλο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να συζητηθεί χωριστά. Χωριστά από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως που γίνονται Μαρτί σήμερα. Πήραμε το μαθήμα μας από το TTIP. Υπάρχουν κάποια ρυθμιστικά θέματα τα οποία δεν κολλάνε σε μια εμπορική συμφωνία. Να, που υπάρχει διαφωνία και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να προσπαθήσουμε να τα βρούμε με τη ΣΥΠΑ τώρα για τον ΠΟΕ και σχετικά με την Κίνα, δύο λόγια. Αυτό που έκανε η Επιτροπή, δηλαδή να ανταποκριθεί σε κάποια αιτήματα, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, το είπε ο κ. Ντεμαρτή. Ότι πρέπει να συνεχίζουμε σε αυτή τη ρότα, γιατί υπάρχει περιθώριο ελιγμών. Έχουν κάποιους ισχυρισμούς βάσιμους νομικής φύσεως σχετικά με το δεύτερο βαθμίο όργανο και την λειτουργία του. Για την Κίνα πολύ σοβαρό, τα λέμε στην μελέτη, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ καλή, συμφωνία, πολύ καλή συνεργασία Ένωσης Ιαπωνίας. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά την Κίνα. Να πάμε για ε, μία, πάμε μία στάση συνολική και για νέα. Ό,τι και να πούμε στην Κίνα θα πρέπει να βλακούν πολύ. είπα δεν είναι πια η στέση να συγκροτήσει κάποιο συνασπισμό γύρω από αυτήν. Να, η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα βάλω μια τελεία και ευχαρίστως να σας ε, απαντήσω ότι ερωτήσεις έχετε. Yeah, thanks a lot. Who will be the first? Oui, euh, je, je vous entends, Monsieur Κύριε Τσέι, σας άκουσα. Μας είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές τακτικές. Άλλες εμείς, άλλες είπα. Ε, βέβαια. Ε, αυτή είναι απότομη, είναι αγρήκη, αλλά αποτελεσματική εμείς φοβόμαστε. Είμαι θα διηρημένοι. Τα είδαμε τους αμέσως προηγούμενους μήνες. Ένα αυτό. Άλλο. Για πες πιο συγκεκριμένα. Να σας παραπέμπω σε αυτά που έχει το website του εμπορικού εκπρόσωπου, τον είπα. Για αυτούς Όλα, όλα είναι υποσυζήτηση, όλα είναι στο τραπέζι. Η γεωργία, η βιομηχανία, ε, τι γίνεται με τα διασυνοριακά δεδομένα. Ε, όχι, δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό είπατε για τη γεωργία. Πιο πολλέ είναι δικέ μας εξαγωγές και όχι εισαγωγές. Αλλά το συμφέρον τους σήμερα, σαφώς, τι είναι να υπάρχει μια ευθυγράμμιση νομοθετική για μας αφόρητη. Για τα μεταλλαγμένα, να τι θέλουν και στο αμερικανικό έγγραφο που διάβασα, μας λέτε ότι υπάρχουν βήματα πρόοδου για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, μα για το COP21 τίποτα, κουβέντα. Ούτε σε αυτό συμφωνούμε. Τι σενάρια έχουμε, τι επιλογές έχουμε. Να μας ακούσουν. Να μας ακούσουν. Δεν θέλουμε TTIP, λένε. Να διαπραγματευτούμε τα ρυθμιστικά, να μην διαπραγματευόμαστε σαν να είναι όλα εντάξει. Ε, να μην είμαστε το κορόιδα της υδρογείου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να παρουσιάσω διάφορες σκέψεις που έχω. Καταρχάς, σε σχέση με τις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι σαφές ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε υπέρ των ε, συμπερασμάτων της ε, διασκέψεως για την καταπολέμηση των κλιματολογικών συνεπειών, των συνεπειών στο κλίμα μάλλον της υπερθέμανσης και των αποφάσεων της συνάντησης κορυφής των Παρισίων. Πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια συμφωνία, ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανικής δραστηριότητας, όταν δεν αναγνωρίζεται η ευθύνη αυτής της δραστηριότητας στην αηφόρο ανάπτυξη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ξεπεραστούν οι διαφορές αυτές. Δεύτερον, σε σχέση με τις ε, αλλαγές στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, όπως επίσης και ε, των διαιτητικών δικαστηρίων, και μετά από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Τρόμπ Εμείς ε, γύρω από όλα αυτά στην Επιτροπή μας έχουμε ε, θα έλεγα συγκεντρώσει την προσοχή μας σε θέματα όπως το Δημόσιο Φόρουμ το οποίο συνοδεύει σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο τις δραστηριότητες του ΠΟΕ. Και στο φόρουμ αυτό εκπροσωπούνται ε, βουλευτές ε, από όλες τις χώρες μέλη του ΠΟΕ. και δεν μπορούν ε, να δεχτούν τις θέσεις τις οποίες προτείνουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα δικαστήρια τα διαιτητικά. Η κατάσταση είναι διαφορετική λοιπόν και οι εμπορικές δραστηριότητες βασίζονται σε συγκεκριμένα θεμέλια και ένα από τα θεμέλια αυτά είναι ακριβώς το Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών καλύτερα. Μας είπατε επίσης ότι στον τομέα της διακανονιστικής συνεργασίας και σχετικά με, τις, ε, με, τους, με τα μη δασμολογικά εμπόδια έχουν υπάρξει κάποια βήματα. και προβλέπεται να γίνουν κάποιες συζητήσεις με διαφορετικό τρόπο από τις συζητήσεις που είχαν συζητηθεί σχετικά με το TTIP. Και συνεχίζουμε μία ακόμα ερώτηση. Το εμπορικό έλλειμμα με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι απλά είναι συνοδευτικό ή είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε άλλους παράγοντες όπως η αποδοτικότητα ή η παραγωγικότητα, το επίπεδο της ζήτησης, της κατανάλωσης. Πολλοί είναι οι Αμερικανοί πολίτες και καταναλωτές οι οποίοι θεωρούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα πιο κατάλληλα για τις ανάγκες τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ε, πώς μπορεί κανείς να δει ε, πού επιρρύπτεται η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Από δική μου πλευρά να κάνω δύο σχόλια. Α, ο κύριος Σόλτς πρώτος. Συνεχίζει ο πρόεδρος. Το θέμα με τις ε, σχέσεις με την Κίνα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα του Τραμπ, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κινηθούμε με στην ίδια κατεύθυνση όπως είπα σε ό,τι αφορά την Κίνα, η συζήτηση που γίνεται με την ε, κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ουσιαστικά η μοναδική προσέγγιση, κοινή προσέγγιση που προέκυψε ήταν σε σχέση με την Κίνα. Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα σε σχέση με το γεγονός ότι φυσικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το εμπορικό πόλεμο αυτό. Θέλω να πω ότι γενικά πιστεύω ότι είναι πιο ανοιχτή και δέχονται πιο πολλές συζητήσεις σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ. Συζητήσεις που να μην είναι και μόνο προς το συμφέρον τους, θεωρώ. Το να προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα τείχο ε, έναντι τη Κίνα. δεν θα είναι και πολύ ωφέλιμο. Σε κάποιε περιπτώσει η προσέγγιση των ΗΠΑ έναντι τη Κίνα. ενδεχομένω να φαίνεται υπερβολική. Αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε κάποιες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του σχετικού σώματος στον ΠΟΕ. Αυτό το αρνούταν διαρκώς ο εκπρόσωπος των είπα. Και με το επιχείρημα, με την τοποθέτηση ότι τους υποστηρίζει η Κίνα. Μα δεν είναι δυνατόν η συζήτηση να γίνεται σε τέτοιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω συνεργασία στη βάση αυτή. Ο κ. Σόλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά μου να θέξω και εγώ δύο πτυχέ, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσω κάποια ζητήματα και να κάνω μία διάκριση. Ποιο είναι τελικά αυτό που ωφελείται από τη νέα αυτή συμφωνία. Και εδώ επαναρχόμαστε πάλι στο ερώτημα και θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την απόψη και την απάντηση ποιοι είναι οι όροι ουσιαστικά παραγωγής, πώς επηρεάζει αυτό το περιβάλλον, πώς επηρεάζει αυτό τα θέματα πολιτικής απασχόλησης, το θέμα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, το θέμα της απασχολησιμότητας και της εμπορευσιμότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Πού είναι ακριβώς αυτή η προστιθέμενη αξία το... της συμφωνίας αυτής. Αλλά το θέμα είναι προφανώς αν είναι εντελώς διαφορετική η τοποθέτηση των δύο εταίρων για την εμπορική πολιτική των δύο πλευρών. Ο καθένας έχει κατά νου κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις καθολικές, τις παγκόσμιες επιπτώσεις αυτές τις αγνοούμε. Άρα, πώς θέλουμε να εξελιχθεί η συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη ενός νέου πολυμερούς προγράμματος. Να μην κοιτάμε δηλαδή μόνο διμερώς το καθαρό όφελος, να κοιτάξουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος και αλλού. Έχουμε μία μελέτη για την αντίκτυπο όλων των ε, συνημένων, ε, συναυθέντων ε, τέτοιων συμφωνιών. θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρξε καμία συνέπεια. ΣΥΤΑ, 7 κτλ. Και ενδεχομένω θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τελικά ουσιαστικό αντίκτυπο ή ο αντίκτυπο που θέλαμε. Ενδεχομένω. Λοιπόν, αυτοί οι διμερεί συμφωνίες να έχουν αντίκτυπο και σε πολυμερέ επίπεδο. γιατί μετά θα έρθουν οι αναδυόμενες οικονομίες και θα λάβουν καθόλου υπόψη τις συνθήκες αυτές. Πώς εκτιμάτε λοιπόν εσείς το θέμα των μεγάλων ε, ομίλων, διεθνικών ομίλων που και η οικονομική, πολιτική και η εμπορική πολιτική των ε, Αμερικανών στην παρούσα φάση είναι τελικά τέτοια που να ακολουθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Πού πιστεύετε λοιπόν την πραγματικά υπεραξία μιας τέτοιας ε, διάταξης, μιας τέτοιας ε, συμφωνίας. Πίτερ. Σας ευχαριστώ πολύ και έχω υπόψη μου ότι δεν έχετε πολύ χρόνο και δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, μία από τις ερωτήσεις που ακούσαμε για τη Γεωργία. Κατά πόσον η Γεωργία θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ή όχι. Και πάλι, Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο διαφορετικών ζητημάτων πρόσβαση στην αγορά και ρυθμιστικά ζητήματα. Είπατε ότι, ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ στην ασφάλεια τροφίμων είναι μη βιώσιμη και είναι κάτι το απευκταίο. Και ακριβώς αυτό λέω, ότι μπορούμε να κοιτάμε τα θέματα τα ρυθμιστικά διαφορετικά σε ό,τι αφορά ξεχωριστά μάλλον σε σχέση με τα ζητήματα πρόσβασης στην αγορά. Το ερώτημα που θέσατε για τη διαφορά μεταξύ της προσέγγισης στο TTIP και εδώ πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να ακολουθήσει να ακολουθηθεί αυτή η οδός. Όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής κ. Δεμαρτή σήμερα το πρωί, πολλές από τις ΜΚΟ είπαν το εξή ότι τα αριθμιστικά ζητήματα δεν έχουν ε, θέση στην εμπορική συμφωνία. Η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να είναι μια συμφωνία για το εμπόριο. Τα αριθμιστικά ζητήματα θα πρέπει να τα επιλύσουν οι, ίδιοι, οι ίδιες ρυθμιστικές αρχές. Για να δούμε κατά πόσον υπάρχει σωστή προστασία για το θέμα της ε, γεωργίας. Στις οδηγίες διαπραγμάτευσης πουθενά δεν διευκρινίζει η κυβέρνηση. Θέλουν να, να ξεφορτωθούν την ευρωπαϊκή προσέγγιση για την βιοτεχνολογία. Λένε, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ ο κόσμο θα πρέπει να γνωρίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ έχει μια καλή πολιτική βάση επιστημονικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα βιοτεχνολογία. 70 έχουν εγκριθεί για την ε, πρόθεση στην αγορά και αυτό βασίζεται στις δικές σας επιστημονικές εκτιμήσεις και έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας και αυτό δεν θα πρέπει αναγκαστικά να μπει στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων, γιατί είναι και θα καταλήξουμε με το θέμα του ΠΟΕ. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε. Το να δημιουργήσουμε ένα τείχος ε, αντίσταση στην Κίνα δεν είναι ενδεχομένω ο πιο έξυπνος τρόπος. Η κινέζικη ηγεσία νομίζω αναγνωρίζει και έχει αναγνωρίσει σε διάφορε περιστάσεις ότι η υπερπαραγωγή που υπάρχει στην οικονομία της αποτελεί ένα, μια ένδειξη ότι η οικονομία δεν λειτουργεί όσο καλά θα έπρεπε. Και θα πρέπει να κάνουμε κάποιε μεταρρυθμίσεις και για του δικού του σκοπού. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υπερπαραγωγικότητα, η υπερπαραγωγή σε, διάφορες, ε, σε διάφορους κλάδες, όχι μόνο στο χάλιβα, αλλά και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω απελευθέρωση κατά την ε, συζήτηση στον κύκλο της Ντόχα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι το εξή, ότι ο υπόλοιπο κόσμος, όχι μόνο η ΕΠΑ, Ούτε μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μόνο η Ιαπωνία, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ουσιαστικά θέλει να σπρώξει την Κίνα να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνει, γιατί αυτή η υπερβολική παραγωγή, οι επιδοτήσεις και το καθεξής, επηρεάζουν και τις Βραζιλιάνους και τους Ευρωπαίους, τους Ονδονήσιους και όλο τον κόσμο. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τμήματος ενός ε, διπλωματικού διαβήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε μέτωπο ενιαίο και κατά της ε, Κίνας. Για το σώμα ε, επίλυσης διαφορών. Ε, πώς λειτουργεί. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ανησυχίε για το σώμα αυτό είναι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ήταν μόνο στην κυβέρνηση Τραμπ το γεγονό ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δαπανίσει τόσο πολύ χρόνο να συζητά τέτοια θέματα για τέτοιε λεπτομέρειε που είναι, διπλωμα... είναι προβληματικέ στα πλαίσια του σώματο επίλυση διαφορών ε, και του πω, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάποια κυβέρνηση αυτή ένα εταίρο που θέλει να εγκαταλείψει το σύστημα. Όχι, δεν θα πολύ χρόνο σε αυτό. Και έτσι πολλά από τα θέματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στι ανακοινώσει Τη Αμερικανικής κυβέρνηση, Η μία διαφορά που πραγματικά υπάρχει μεταξύ της ε, Αμερικανικής κυβέρνηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, δασμούς. Καθορισμό των προστήμων σε ό,τι αφορά τους ε, τελωνιακούς δασμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάει και διδάξουμε πρώτα την διαδικασία. Η κυβέρνηση θα πρέπει να τα εξετάσει αυτά, γιατί χωρίς το σώμα επίλυσης διαφορών η κατάσταση θα δυσκολέψει. Και αυτό μας οδηγεί στο τελευταίο ερώτημα, φαντάζομαι, του κυρίου Σόλτσα για την προστιθέμενη αξία σε μια διμερή συμφωνία και κατά πόσον ε, οι διμερεί συμφωνίε ουσιαστικά βλάπτουν το πολυμερέ επίπεδο. Νομίζω ότι όλοι θα προτιμούσαμε το πολυμερέ επίπεδο και πολλέ χώρε που συμμετείχαν στο γύρο τη Ντόχα τόνισαν ότι πολλέ αναδυόμενες οικονομίε δεν ήθελαν να προβούν σε απελευθέρωση περαιτέρω ε, αν η Κίνα δεν ε, περιόριζε την παραγωγή τη. Και εδώ λοιπόν αυτό είναι ακόμα ένα επιχείρημα για το οποίο η Κίνα θα ωφελούταν από την μεταρρύθμιση της παραγωγής της. Χωρίς αυτή, τα μέλη του γύρω της Δόχα, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προέβαιναν πολύ απλά σε διμερείς συμφωνίες. Και όπως είπατε, αυτές οι διμερείς συμφωνίες έχουν και θετικό αντίκτυπο στο πολυμερές επίπεδο. Έχω πολλά ακόμα να συζητήσω, αλλά νομίζω ότι καλά θα κάνω να σταματήσω στο σημείο αυτό. Γιατί δεν ε, προλαβαίνετε κιόλα με το χρονοδιάγραμμά σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Είμαι πεισμένο ότι η συζήτηση για τι ευρωπαϊκές Εμπορικέ σχέσεις και τον αντίκτυπο για τον ΠΟΕ θα επανέλθει εδώ πολλέ φορές. Και φυσικά, Πίτερ, είμαι βέβαιο ότι θα στραφούμε και πάλι προ εσά για να διδαχτούμε από την εμπειρία σας. Σα ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 14 στην ημερησία διάταξη και έτσι σε πέντε λεπτά θα περάσουμε στο σημείο 15 που αποτελεί μια ακρόαση για την ευρωπαϊκή και ασυντική συνδεσιμότητα και ποιος είναι αντίκτυπος του εμπορίου. Okay.

Υπότιτλοι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 Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Μάλιστα, συνάδελφοι, πάμε στο 15 της ημερήσιας διαταξής. Η δημόσια ακρόαση, λοιπόν, για τη συνδεσιμότητα Ευρώπης-Ασίας. Είμαι πεπισμένος ότι το θέμα αυτό είναι ενδιαφέρον αλλά περίπλοκο λόγω της φύσης της συνδεσιμότητας καταρχάς που δεν είναι κάτι το οποίο ορίζεται πάρα πολύ επακριβώς αλλά επίσης λόγω και της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στις δύο ε, περιοχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν δημοσιεύσει ένα κοινό έγγραφο το οποίο ονομάζεται Connecting Europe and Asia. Σημείο εκκίνησης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Και έχουν ήδη καταθέσει ορισμένες προτάσεις. Από την άλλη, Και η Κίνα έχει προσπαθήσει να κάνει κάποια τέτοια βήματα. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στα πλαίσια της κινέζικης στρατηγικής το ερώτημα το οποίο τίθεται βέβαια είναι αν οι δύο στρατηγικές αυτές είναι συμπληρωματικές ή ε, δημιουργούν προβλήματα η μία στην άλλη. και σε ποιο βαθμό ε, οι διευκολύνσεις που μπορεί να υπάρξουν στον τομέα αυτό θα είναι δημιουργίες επενδύσεων και σε ποιο βαθμό είμαστε σε θέση να πιέσουμε την Κίνα ε, και κατά πόσον η Κίνα θα κυριαρχήσει πλήρως στον τομέα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα ενδιαφέροντα, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις στρατηγικής φύσεως κάτω από τον τίτλο αυτό Europe-Asia Connectivity. Για να τα συζητήσουμε αυτά όλα. Έχουμε εκλεκτούς εμπειρογνώμονες μεταξύ μας Ελπίζω να είναι ζωηρή η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Έχουμε λοιπόν αρκετούς και εκλεκτούς εμπειρογνώμονες θα διευθύνουν την συζήτηση κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες και όχι εγώ. Η Γιάννα έχει λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που θα μπορέσω να διευθύνω τη συζήτηση ενός θέματος το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας για πάρα πολλά. Τι είναι το Borderlec λοιπόν είναι μια σειρά δημοσιεύσεων για την εμπορική ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική ομάδα που ασχολείται με θέματα δίκαιου εμπορίου Γενικά τα θέματα του εμπορίου βέβαια συζητιούνται σε, περίπτωση, σε επίπεδο κυρίως επιτροπών του Συμβουλίου κτλ. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει η συνδεσιμότητα στην εμπορική δραστηριότητα. Καταρχάς, η στρατηγική των Κινέζων, τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κατανοηθεί επίσης και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύθηκε το, το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά θα έχουμε κάποιες κατά περίπτωση μελέτες για το πώς η συνδεσιμότητα αυτή είναι γεγονός, λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καλά σε σχέση με θέματα εργασιακά, σε σχέση με θέματα ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε πολλούς και ενδιαφέροντες ε, ομιλητές. Θα ήθελα να ζητήσω το πρώτο πάνελ να προετοιμαστεί δεν χρειάζεται να ανέβουν στο βήμα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τις ομιλίες του πρώτου πάνελ να κατανοήσουμε την στρατηγική των Κινέζων, να δούμε σε ποια επίπεδα βρίσκονται οι διαφορές ανάμεσα στην Κίνα και στην Ευρώπη. Ο πρώτος ομιλητής είναι εμπειρογνώμονας για τα θέματα της διεθνούς πολιτικής της Κίνας με το Ινστιτούτο Μοντένια, ο Τόμας Έντα. Είναι επίσης εκπρόσωπος του Μέριξ Institute. Έχουμε την Άστριντ Κούμαν, στο Γερμανικό Σώμα Συνεργασίας για την Ανάπτυξη και έχουμε και τον κύριο Βαϊόλα ο οποίος είναι οικονομικός σύμβουλος στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για θέματα αναπτυξιακά στην Νοτιοανατολική Ασία. Και έχουμε και τον κύριο Wei Shi, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού Εμπορίου στην Πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Έχουμε και τον Φρανσουά Γκοντμαν. Εν πάση περιπτώσει όλοι οι ομιλητές θα κάνουν μια πολύ σύντομη εισαγωγική παρέμβαση και μετά θα ξεκινήσουμε ερωταπαντήσεις για 20-25 λεπτά. Φανσουά Ευχαριστώ Γιάννα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να φανώ ρεαλιστής και όχι σκεπτικιστής, αν και θα πρέπει να πω ότι μην χάσετε τον ύπνο σας για τη συνδεσιμότητα και για την Κινέζικη Πρωτοβουλία. Ε, η συνδεσιμότητα είναι θα έλεγα μια λέξη παγίδα στην ουσία. Μπορεί να είναι τα πάντα αλλά μπορεί να είναι και τίποτα ταυτόχρονα. Όλα συνδέονται ακόμα και οι φωτογραφίες μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή εξετάσει κανείς το εξαιρετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το σημαντικό εδώ είναι οι προσπάθειες τις οποίες κάνουν για μεγαλύτερη εξιστρέφεια οι Κινέζοι στον τομέα των ψηφιακό και στον τομέα των επικοινωνιακών ε, με τη νέα αυτή στρατηγική, το νέο αυτό δρόμο της Κίνας προς τα έξω. Είναι μια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει ενδιαφέρον όχι μόνο από το 19ο αιώνα αλλά πολύ παλιότερα και μια ιδέα επίσης ε, την οποία είχε προωθήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεκαετία του, ε, του 90 Πρόκειται λοιπόν για τη στρατηγική που ονομάζουμε BRI. Είναι πολλά τα στοιχεία της πολιτικής αυτής, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει κιόλας η πολιτική αυτή συνολικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλευρές στρατηγικής, τα οποία πολλές φορές, ε, οι οποίες πολλές φορές ε, μας απασχολούν, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα πολλές φορές εξαφανίζονται τα πάντα και με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι Κινέζοι με έναν χαοτικό τρόπο, με έναν μαζικό τρόπο κάποια συνθήματα ακούγονται πάρα πολύ δυνατά, επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν, κάποια άλλα συνθήματα εκεί που ακούγονται χάνονται. Και γι' αυτό όταν βλέπετε τους επίσημους κινέζικους αριθμούς όχι αριθμούς ε, οι οποίοι μπορεί να ε, δοθούν σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών, θα δείτε ότι αυτά ε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία λέγουν. Το 2014 η Κεντρική Τράπεζα έλεγε ότι θα διαθέσει στα πλαίσια της χρηματοδότησης αυτής της στρατηγικής το 1 τέταρτο σχεδόν των αποθεματικών των συναλλαγματικών της χώρας. Όταν βλέπετε όμως το τι πραγματικά ξοδεύουν. Άλλοι λένε ότι ξοδεύουν 14 δις το χρόνο, άλλοι λέγουν ότι ξοδεύουν 25 δις, άλλοι λένε ότι είναι από 150 σε 250. Φυσικά πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ξοδεύει η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά όχι αυτά τα τρεις τα οποία κάποτε λέγαμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας οι Ιάπωνες δημιουργούν περισσότερες υποδομές στον τομέα από ότι οι Κινέζοι στην Νοτιοανατολική Ασία συνολικά. Υπάρχουν πολύ περισσότερες επενδύσεις των Ιαπώνων και των Κορεατών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξαιρώντας τα Βαλκάνια που είναι ειδική περίπτωση. Συνεπώς λοιπόν η διαφήμιση πολύ ε, έκανε τη δουλειά της, Υπάρχει βέβαια και κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην Κίνα γιατί α, κατηγορείται η Κίνα ότι ήταν ιδιαίτερα κυριαρχική στις προτάσεις τις οποίες κάνει, υπεριαλιστική σχεδόν και γι' αυτό πολλές φορές έπεσαν στην ίδια τους την παγίδα και άλλοι έχουν πέσει όμως σε παγίδες. Σήμερα σαν παράδειγμα διαγράφονται για πρώτη φορά από την Κίνα χρέη σε σχέση με την στρατηγική αυτή. Είναι κάτι το οποίο είχε ανακοινωθεί εν μέρη ε, στα πλαίσια του τελευταίου ΦΟΚΑΚ, της κορυφής δηλαδή ανάμεσα στην Αφρική και την Κίνα και αυτό δείχνει το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της ίδιας της στρατηγικής την οποία ακολουθεί στον τομέα των επενδύσεων η Κίνα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ βιώσιμη από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή, πάντως το BRI είναι και μύθος και δεν υπάρχει. Είναι οικονομικά κάτι το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Υπάρχει ένας ειδικό εμπειρογνώμων στο Πανεπιστήμιο εδώ των Βρυξελών που έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο λέγοντας ότι ναι μεν θέλει να φτιάξει υποδομές λιμενικές, αεροπορικές, ιδεοδρομικές... αυτά που κάνουν καλά οι Κινέζοι μαζί με την ψηφιακή ε, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικές πληρωμές. Υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο έχει σχέση με τον BRI, είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Όλοι επηρεάζονται από αυτή την πρωτοβουλία αλλά κάποια περάσματα τα οποία υπάρχουν όχι σε επίπεδο θαλάσσια μεταφορών, υπάρχουν κάποια περάσματα εμπορικά στα οποία οι Κινέζοι προσπαθούν να ενισχύσουν την παρουσία τους να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια διεύρυνση των, ε, της γεωμετρίας της εσωτερική τους ανάπτυξης και οικονομίας και ποσοτικά δεν είναι παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των επενδύσεων της Κίνας και της κατανάλωσης. Βλέπετε χάλιβας, ε, ίαλος, χαλκός. Το 90% είναι αυστηρά εσωτερικές παραγωγές για εσωτερικές ανάγκες. Όμως η Κίνα ταυτόχρονα λειτουργεί με κανόνες ή και χωρίς κανόνες, αλλά οι κανόνες όταν υπάρχουν είναι εντελώς διαφορετικοί από τους δικούς μας. Και εμείς κάποτε δεν είχαμε και πάρα πολλούς κανόνες, η συνένεση για διεθνείς κανόνες εμφανίστηκε για κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες, ιδιαίτερα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΣΑ και τα λοιπά τα τελευταία χρόνια. Η βασική πρόκληση λοιπόν για την Ευρώπη είναι το εάν θα μείνουμε ικανοποιημένοι ε, μένοντας στην δική μας εσωστρέφεια με τους δικούς μας κανόνες, με τα δικά μας προγράμματα τα οποία είναι βιώσιμα και να βλέπουμε την Κίνα να κατακτάμε τον υπόλοιπο κόσμο. Και υπάρχουν πολλές χώρες βέβαια οι οποίες δεν μπορούν να σεβαστούν αυτούς τους κανόνες, δεν μπορούν να είναι αντίστοιχα βιώσιμες οι πολιτικές τους, να προσπαθούν ε, να προσαρμόσουν τους Κινέζους στις δικές τους προοπτικές. Οι Κινέζοι θέλουν βέβαια αηφόρα προγράμματα με κανόνες και επιστροφή των επενδύσεών τους και όχι τόσο να είναι βιαστικές επενδύσεις σε άγνωστα εδάφη χωρίς εγγυημένη απόδοση. Ευχαριστούμε και το μα σα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή που μου δίνει την τιμή να πάρω το λόγο εδώ μπροστά σα σήμερα για να σα παρουσιάσω μια άλλη άποψη για το θέμα αυτό και μα ζητήθηκα να μας να μιλήσουμε για τι συγκλήσει και τι αποκλήσει ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή και την κινέζικη προσέγγιση. Να ξεκινήσω με τα βασικά θέματα απόκλησης και στο τέλο θα αναφερθώ στα πιο σύντομα θέματα σύγκληση. Να σα πω δύο λόγια καταρχά, να σα πω ένα μικρό περιστατικό σε ό,τι αφορά μια βάση δεδομένων που οικοδομήσαμε στο Βερολίνο να περιλαμβάνει πλέον 1500 έργα σε ό,τι αφορά τέτοιε πρωτοβουλίε. Καταρχάς, λοιπόν, να σα πω την ιστορία. Το 2017 ήμουν σε ένα workshop σε μια ημερίδα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ε, επιστήμονες αλλά και Κινέζους εκπροσώπους. Ε, υπήρχε λοιπόν μια συνήθιση συζήτηση για το τι ακριβώ είναι το BRI. Ο επικεφαλή τη κινέζικη αντιπροσωπεία ε, σηκώθηκε και είπε ότι το EBRI είναι η παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό. Ε, τι σημαίνει ακριβώ αυτό, Η απάντηση προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Βιωσιμότητα. Τι σημαίνει λοιπόν πάλι αυτό, εξήγησε περαιτέρω ότι η παγκοσμιοποίηση δική σα δεν είναι βιώσιμη. Κοιτάξτε τον Τραμπ, κοιτάξτε τον Brexit. Η δική μα παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη για μας. Ποιο είναι φυσικά εμά, ε, Φυσικά αυτό είναι η Κινέζικη, το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα και γι' αυτό είναι το πρίσμα υπό τον οποίο θα πρέπει να κοιτάξετε την πρωτοβουλία BRA. Η στρατηγική για την σύνδεση Ευρώπης και Ασίας που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και βιωσιμότητα και μια συνδεσιμότητα βάσει κανόνων. Αυτό που δεν προκαλεί έκπληξη σε σχέση με τον περιστατικό που σα ανέφερα είναι ότι είναι διαφορετικέ αντιλήψει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόθεση του BRI είναι να δημιουργήσει νομιμότητα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, μεταξύ άλλων με οικονομική ανάπτυξη, να δοθούν συμβάσει στι κινέζικε εταιρείε και θέσει απασχόληση στου Κινέζου πολίτε. Όταν κοιτάμε τα κινέζικα project στη βάση δεδομένων μας και εδώ πέρα έχουμε κάποιες ε, από τις περιπτώσεις αυτές στους χάρτες μας. Φυσικά, οι κινέζικες εταιρείε ε, κερδίζουν τις πιο πολλές ε, συμβάσεις και γι' αυτό τα πανάλογα και εκείνα τα χρήματα. Όταν εξαιρούμε τους ανοιχτέ και διαφανείς ε, διαδικασίε, ε, αυτοί θα κερδίζουν. Γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι τα πιο πολλά project είναι αρκετά χαλαρά σε ό,τι αφορά τι ρυθμίσει για το περιβάλλον. Και έτσι φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη ε, φροντίδα σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα. Κάποιε και μικρέ και ευάλωτε οικονομίε έχουν πάρει δάνεια. Ακόμα και είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσουν να τα ξεπληρώσουν αυτά. Και κοιτώντα διάφορα προγράμματα για οικοδομέ, σε ό,τι αφορά το BRI. Βλέπουμε τα θέματα περιβαλλοντική ε, βιωσιμότητα. Οι κινέζικε δαπάνε ε, στην Ευρώπη έχουν επικεντρωθεί στα Δυτικά Βαλκάνια σε ό,τι αφορά ε, μέρη δίπλα σε ε, αυτοκινητόδρομους και κυρίως σε για παραγωγή ενέργεια από ορυκτά καύσιμα η χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα και από τι ευρωπαϊκέ πηγέ έχει στεγνώσει πλέον. Η Κίνα λοιπόν έχει δει το άνοιγμα και βοηθά τι εταιρείε τη να αντικαταστήσουν τη μειωμένη ζήτηση που έχει στην Κίνα. Ένα βασικό στόχο λοιπόν είναι να υπάρχουν κινέζικε εταιρείε σε διάφορου τομεί, στην μεταφορέ, στην ενέργεια, ψηφιακό, ε, στι τηλεπικοινωνίε και να αναδεχθούν σε παγκόσμιε ηγέτε. Και υποτίθεται ότι θα βρουν στην περίπτωση αυτή από μια θέση ισχύω. Θέλουν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με σωστούς ε, όρους και να είναι πιο ανταγωνιστικές χωρίς να εξαρτώνται σε χρηματοδότηση από κρατικέ τράπεζε, προκειμένου να μπορέσουν να εγκαθατρήσουν τη θέση του στο μακροπρόθεσμα. Προτού όμω ε, κλείσω, να αναφέρω άλλο ένα θέμα απόκληση για ένα πιο μικρό τμήμα του BRI. Τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται, από την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και την IIIB και η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να επεκτείνουν και να διευρύνουν την συνδεσιμότητά τους και στην παρούσα φάση πέρα και από άλλους στόχους από αυτούς που ανέφερα για την Κίνα. Αυτό καταδεικνύει και ένα περιστατικό για την επικοδομητική συνεργασία το οποίο θέλω να το αναφέρω. Ε, ο αγωγός ε, Trans Όταν ξεκίνησε η χρηματοδότηση, όταν ε, γίνεται από πολυμερές σε πολυμερές επίπεδο, όπως το WB, EBRD και ETEP και AIIB, τότε ένα έργο δεν μπορεί να ακολουθήσει το μοντέλο που σας ανέφερα προηγουμένως με τις <coughs> χρηματοδοτήσει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στην τήρηση των προτύπων και μια διαφανή διαδικασία με ίση πρόσβαση για ευρωπαϊκέ εταιρείε. Και μια περαιτέρω συνεργασία από την έννοια αυτή θα μπορούμε να πούμε ότι συμμορφώνεται και με την επέκταση του TNT και με τους, τα σχέδια διαδρόμων BRI. Και έτσι λοιπόν ένα, μια επικεντρώση λογική θα ήταν και η Μαύρη Θάλασσα, η οξύνη πόντο, η Βουλγαρία, η Ρωμανία, η Ουκρανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κούμαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τιμή μου να συμμετέχω και να σας πω τις απόψεις μου για το PRI. Έχω πήρα 15 ετών για αυτή την υπόθεση. Βεβαίω και έχουμε την οπτική γωνία τη Ευρώπη, αλλά μιλούμε τώρα για συνεργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε τον BRI, να καταλάβουμε όμως και την οπτική γωνία της άλλης πλευράς. Πέρασαν τόσα χρόνια για να μπορέσει να καταλάβει η Ευρώπη τον BRI για να μπορέσει να απαντήσει μετά το ξεκίνημα στην Αστάνα το 2013 αυτή τη υπόθεση και ε, πήραν κάποιο χρόνο στους Ευρωπαίου ε, να ε, μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την περιέργεια, την σύγχυση, τον προβληματισμό, την παρακολούθηση δηλαδή αυτή τη ε, κινέζικης περιπέτειας του, του, που την ξεκίνησαν οι Κινέζοι το 2013. Για να δούμε, να το απομυθοποιήσουμε λίγο. Να δούμε Τρία θεματάκια βασικά. Πρώτα πρώτα έχουμε αυτό που θα ονόμαζα ε, παρεξηγήσεις σε σχέση με το BRI. Μετά έχουμε κάποια βασικά σημεία για το πώς διαρθρώνεται, πώς λειτουργεί το BRI και επίσης για να δούμε για τη βιωσιμότητα αυτού. Ίσως βρούμε πολλά κοινά που έχουν σχέση δηλαδή με την στατική της ε, συνδεσιμότητας και αυτά ωφελούν και για το να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει δύο σήματα. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμείς το βλέπουμε με κριτική ματιά, θεωρούμε ότι είναι απλώς ε, ένα σλόγγαν, ότι είναι πράγμα κινέζικο εισαγωγικά, κομμουνιστικό, ότι δεν είναι πλάνο, ε, ότι θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια παγκοσμιοποίηση παράλληλη στην ε, υπάρχουσα. υπερπαραγωγή, όπως είδαμε να γίνει σε πολλά μέτωπα φέτος, τσιμέντο και χάλιβας. Λοιπόν, αυτά τα λέμε μεν, αλλά περιέχουν και κάποιες παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Το 75 με 80% των έργων που χρηματοδοτούνται από όλες τις αναπτυξιακές τράπεζες και FW τη η Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξη πάνε στη Γερμανία και στην Ευρώπη, στι επιχειρήσει. Τα είναι αυτά στη συνέχεια από τον κύριο Σέντερ προηγουμένω. Για να δούμε τώρα κάποια βασικά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ε, δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι γίνεται με αυτή τη στρατηγική. Είναι περίπλοκο. Μπλέκει πολλές περιφέρειες, μπλέκει πολλές χώρες δεν έχει να κάνει μόνο με έναν φορέα, έναν οργανισμό, ούτε στην κοινότητα πουθενά άλλο. Γι' αυτό και μας δημιουργεί μια σύγχυση. ...130 μνημόνια και υπομνήματα, συμφωνίες, προγράμματα, διάφορα πλαίσια για να καλύψουν τις τρεις διαστάσεις συνδεσιμότητας που αναδύονται από αυτό το concept BRI του 15. Είναι κάτι που προέκυψε από, την, από το Υπουργείο Εμπορίου, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την Αρμόδια Εμπορική Επιτροπή και έχουν εκδώσει ένα σωρό ανακοινοθέντα από το 2013 ε, ενέργεια, συνεργασία, περιβάλλον, προγράμματα δράσης και πολλά άλλα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από φορείς, όχι μόνο κινέζικους, αλλά πραγματικά αυθεντικά διεθνείς. Ένα σώρο think tank, οργανισμούς που ασχολούνται με το BRI. Άρα, δεν υπάρχει ένας ε, ούτως είπε αποδέκτης ενός τηλεφωνήματος στο Πεκίνο για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει ένας φορέας που το διαχειρίζεται και έχουμε ένα σωρό διάφορους θεσμούς, διάφορες αμψιακές τράπεζες, διάφορους μη κινηζικούς φορείς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε πάνω από 25 διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και όχι μόνο που συνδέονται με πρωτοβουλίες, με συμπράξεις, προγράμματα και υπάρχει και το θεματολόγιο του 2030. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων ε, των αναπτυξιακών, των στρατηγικών Δικαίως προβληματιζόμαστε, θα δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι αντιπαραγωγικό αυτό το θέμα για το θεματολόγιο. Καθαρή ενέργεια, αποτελεσματικά δίκτυα. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε το ότι αν δεν προστατευτεί και το περιβάλλον θα πρόκειται για ένα ναυάγιο. Οπότε έχουμε έργα υποδομής, πολλές ε, επενδύσεις, ε, βλέπω εδώ πέρα μεγάλες ε, ευκαιρίες. Έτσι θα πρέπει να δούμε το θέμα. Όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει κοινό έδαφος να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έργα για να βοηθήσουμε το θεματολόγιο του 2030. Οπότε έχουμε αυτή τη στατική του 2018 του Σεπτεμβρίου για την συνεσιμότητα. αμοιβιότητα, ισότητα όπλων, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να βρούμε τον κοινό παρανομαστή, το κοινό έδαφος, να δυναμώσουμε τις σχέσεις και τους δεσμούς μας με την Ασία, να έχουμε περισσότερη βιωσιμότητα, να πετύχουμε περισσότερα. Και ο έχει το λόγο. Να δούμε τα πράγματα που έχουν των Κινέζων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Πρόεδρο, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής και είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να συμμετέχω σε αυτή την ε, κοινή ακρόαση. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταία τρία χρόνια πριν να ε, ε, έρθω στις Βρυξέλλες εργάστηκα Ω επικεφαλή του τμήματο PRI στο Υπουργείο Εξωτερικών τα τελευταία δύο χρόνια έχω συμμετέχει σε διάφορε συζητήσει σε διάφορα φόρα και είχα ακούσει πολλέ προτάσει σε ό,τι αφορά το BRI. Ε, άκουσα και πολλά εχθρικά σχόλια και πολλές υποψίε, καχύποπτα σχόλια. Πιστεύω ότι είμαι προσωπικά υπέρ του, της πρωτοβουλίας BRI. Έξι χρονών είναι πλέον αυτή η πρωτοβουλία και είναι σημαντική λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή. Αυτό το εξάχρονο λοιπόν παιδί θεωρώ πλέον ότι σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις αξίζει την κριτική που το απευθύνεται, αλλά πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή θα σημαίνει επιτυχία για όλο τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση προετοιμάστηκα λοιπόν στη σημερινή, για τη σημερινή συνεδρίαση και Είδα τα απορίσματα της Διεθνούς ε, Συνόδου για τα τέτοια θέματα στο Πεκίνο πέρσι. πρόκειται λοιπόν για μια τέτοια πρώτη πρωτοβουλία. Και γιατί επιλέξαμε την πρωτοβουλία αυτή. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλό για τη δημοσιότητα. Θέλουμε να υπάρχει διεθνής χαρακτήρας. Θέλουμε να προβληθεί έτσι ως διεθνή πρωτοβουλία, διαφανής πρωτοβουλία. Να είναι λοιπόν ανοιχτή και διαφανή ως πρωτοβουλία. Αυτό ακολουθήσαμε ως πνεύμα και ακούσαμε και άλλες σημαντικές ιδέες για τη μεταρρύθμιση των BRI. Και πάντα εκτιμώ τις προτάσεις αυτές. Δύο τμήματα λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω σήμερα. Το θέμα είναι λοιπόν καταρχάς το σημείο εκκίνησης. από πού ξεκινάει η πρωτοβουλία BRI και γιατί ε, την πρόθεσε η Κίνα, γιατί στην ε, φάση αυτή συγκεκριμένα. Και δεύτερον, να κατανοήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Στο πρώτο τμήμα λοιπόν, γιατί η Κίνα και γιατί τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια συνέχιση του δρόμου του μεταξιού της ε, ιστορίας. Η ιστορία θεωρώ είναι πολύ βασική εδώ. Πολλοί περιγράφουν την πρωτοβουλία BRI ως μία από τις πιο σημαντικές, την πιο σημαντική πρωτοβουλία που παίρνει η Κίνα. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει τόσο μεγάλη πρωτοβουλία η Κίνα. Και γιατί. Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε το ιστορικό παρελθόν. Γιατί Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο δρόμος του μεταξιού της Ασίας ήταν μια πρώτη μορφή παγκοσμιοποίησης. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό υπόβαθρο της παρούσας πρότασης. Κοιτάμε την συνδεσιμότητα, θέλουμε μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ Ασίας και Αφρικής και Ευρώπης. Θέλουμε να υπάρχει συγχρονισμένη αλυσίδα παραγωγής και αξίας. Θέλουμε οι περίκλειστες χώρες να συνδεθούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα υπέβαλε ένα σχέδιο πέρα από τα θέματα αυτά σε επίπεδο οικονομίας. Δεύτερος λόγος, το θέμα της διαδικασία ανοίγματο της οικονομίας. Εκείνα, λοιπόν προτείνει αυτή την ε, πρωτοβουλία αυτή φυσικά και έχει τα συμφέροντά τη η Κίνα. Είμαστε ήδη η πρώτη οικονομία στον κόσμο και είμαστε ο μεγαλύτερο ε, εμπορικό εταίρο για 130 χώρε και περιμένουμε ότι θα είμαστε και η πιο μεγάλη αγορά κατανάλωση σύντομα. Αλλά ακόμα έχουμε το πρόβλημα ε, ότι έχουμε πολλέ ανισορροπίε. Κοιτώντα για παράδειγμα τι δυτικέ επαρχίε τη Κίνα, 72% ε, των εδαφών τη Κίνα, 27% του πληθυσμού αλλά το ΑΕΠ των δυτικών ε, επαρχιών καλύπτει το 20% των, ε, του ΑΕΠ της Κίνας και το 7% των μελαταπών επενδύσεων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τις δυτικές αυτές επαρχίες. Θέλουμε οι δυτικές αυτές περιοχές να αναδεχθούν σε ηγέτη για την μεταρρύθμιση της Κίνας και για τη μετάβαση της Κίνας στο επόμενο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν εστιαζόμαστε στο NDRC και ακριβώς το αρχηγείο, αν θέλετε, το επίκεντρο για τα θέματα αυτά είναι στις δυτικές επαρχίες. Αυτή είναι η εξήγηση της Κίνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτή και νομίζω ότι αυτό δίνει νέα όθηση στην αγορά. Θέλουμε να προωθήσουμε μια ανοιχτή οικονομία. Όλοι γνωρίζουν την αρχή των ε, διαβουλεύσεων, των κοινών ε, κατασκευών και του κοινού συμφέροντος. Αυτό είναι στον πυρήνα της πρωτοβουλίας μας και πιστεύω ότι τελικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εναρμόνιση, ανοιχτή εναρμόνιση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εντελώς νέο σχήμα κανόνων, κάτι που δεν υπάρχει πριν. Όχι, ποτέ δεν ήταν αυτό η πρόθεσή μας. Και να περάσω λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Έχω ένα κατάλογο αριθμητικών στοιχείων και δεδομένων για να σας εξηγήσω από πού προέρχεται, προέρχεται η επιτυχία της Κίνας ό,τι αφορά και την πρωτοβουλία BRI. Και στο δεύτερο τμήμα να κατανοήσουμε τρεις λέξεις κλειδιά σε ό,τι αφορά τον BRI από διάφορα στοιχεία, από διάφορες ε, πλευρές. Καταρχάς, ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Γιατί, Γιατί πρόκειται μια πρωτοβουλία που είναι κοινή σε ό,τι αφορά τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες στον πυρήνα βρίσκεται η ανάπτυξη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, δεν είναι κάτι το σταθερό, το αμετάβλητο. Αν θέλετε να συγκρίνετε με αυτά που προτείναμε στο πρώτο επίπεδο, στην πρώτη φάση του BRI και τώρα τι προτείνουμε, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά υπό εξέλιξη. Και αυτό είναι λογικό άλλωστε γιατί όλα ε, αλλάζουν και εξελίσσονται μέρα με τη μέρα. Δεύτερο στοιχείο, το θέμα της συνδεσιμότητας. Ε, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι πανελίστες. Θέλουμε λοιπόν να εστιαστούμε πιο πολύ σε τέτοια σημαντικά θέματα συνδεσιμότητας. Από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης δημοσιεύτηκε μία μελέτη για την ε, ε, τον χάρτη της παγκόσμιας συνδεσιμότητας και πιστεύω ότι η πρωτοβουλία BRI ουσιαστικά αποτυπώνει τις επιθυμίες αυτές για να υπάρχει μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε ό,τι αφορά τους πέντε πυλώνες για τις πολιτικές, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, τις επιχειρήσεις, πολιτικές και του καθεξής. Τρίτη έννοια τώρα, τρίτο στοιχείο, είναι τα υψηλά πρότυπα, υψηλή ποιότητα και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων. Βλέπουμε τη μετάβαση από τις χρυσές ε, αυτές το μέσα από τις αρχές αυτές. Βλέπετε λοιπόν ε, πως υπάρχει εξέλιξη. Κάποιοι διατείνονται ότι τα προγράμματα, τα έργα της Κίνας δεν είναι τόσο διαφανή και ότι πάντα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εδώ δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα στοιχεία στέκουν. Και αν κοιτάξουμε διεθνή στοιχεία, πέρσι 22 έργα ε, κατανεμήθηκαν, τα μισά από αυτά ήταν από την Κίνα. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, ακολουθούμε μια πολιτική που είναι φιλική προς το περιβάλλον, προς το κλίμα, είναι διαφανής και αμερόληπτη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πλαίσιο αυτό τη συνδεσιμότητα, εξ αρχή ε, διευκρινίσαμε ότι υπάρχουν καλέ ευκαιρίε για να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα μεταξύ των δύο πρωτοβουλειών και έγιναν κάποιε συζητήσει ε, για τα θέματα αυτά. Και υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτέ οι δύο πρωτοβουλίε θα αποφέρουν πιο από τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σα ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η υπηρεσία εξωτερική δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στα θέματα της συνδεσιμότητας. Είναι χρήσιμο νομίζω γιατί δείχνει ακριβώς τις δράσεις που έχω συμπεριλάβει, που έχω συμπεριλάβει στις πρωτοβουλίες αυτές. Είναι η πολιτική δικτύων θα την ονόμαζα, που επιτρέπει τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, των ψηφιακών δικτύων και της ανθρώπινης συνδεσιμότητας. Η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναγνωρίζει τη σημασία της συνδετιμότητας με την Κίνα και με την Ασία γενικότερα και αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρχει μια συνοχή ε, με ε, τις αντίστοιχες πολιτικές της Κίνας. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2018 και τα συμπερόσματα που ακολούθησαν ήσαν έτοιμα τον Οκτώβριο 18 και 19 ε, στη συνάντηση κορυφής του, Ασενά, του ΑΣΕΑΝ. Έχω έξι διαφάνειας για σας εδώ, θα είμαι σύντομος. Οι έξι αυτές διαφάνειες αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα της στρατηγικής και θα υπάρξει και μία διαφάνεια για τα συμπεράσματα. Καταρχάς η σημασία της Ασίας στον εμπορικό τομέα. Η Ασία είναι το 60% του πληθυσμού του κόσμου, 35% των εξαγωγών μας και 32% των εισαγωγών. Επίσης υπάρχει τεράστια ανάγκη για επενδύσεις και υποδομές στην Ασία. Πιστεύουν ότι απαιτείται σε αιτήσια βάση 1,33 επενδύσεων και αυτό αφορά και στην Ευρώπη και τις υπόλοιπες εταιρείες, ε, μάλλον υπήρους και εταιρείες από διάφορες υπήρους. Αυτό δημιουργεί ροές, αυτό δημιουργεί αλληλοεξαρτήσεις και γι' αυτό η συνδεσιμότητα έχει συνέπειες στο πολιτικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή δημιουργήθηκε σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο υπήρχαν εθνικού τύπου πολιτικές, όχι μόνο η Κίνα με τη στρατηγική της, αλλά η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, που έχουν δικές τους ανεξάρτητες στρατηγικές συνδεσιμότητας για τη λεκάνη του Ειρηνικού. Υπάρχει και το πρόγραμμα συνδεσιμότητας του ΑΣΕΑΝ και η Κεντρική Ασία επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. Το μήνυμά μας είναι ένα. Εμείς θέλουμε να συνδεθούμε με τις πρωτοβουλίες αυτές να εμείνουμε σε θέματα ευημερίας γενικά του πληθυσμού αλλά κυρίως βιωσιμότητας και συνεργασίας. Οι στρατηγικές βασίζονται ε, σε δύο κυρίως θέματα. Το θέμα της αηφορίας περιλαμβάνει το περιβάλλον, την οικονομική αηφορία και βιωσιμότητα δημοσιονομικά θέματα και κοινωνικά θέματα. Αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας συζήτησης που αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συνδεσιμότητας. Και τίθεται το θέμα φυσικά και της υπερχρέωσης και τα κοινωνικά επίπεδα προστασίας. Η στάση που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα είναι ε, θα έλεγα σφαιρική, καλύπτουμε όλους τους τομείς και τους πολίτες και ε, τις επικοινωνίες και τις μεταφορές <clears throat> και τα ψηφιακά θέματα δημιουργώντας ένα, επιδιώκοντας τη δημιουργία πολυμερούς περιβάλλοντος που διέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες. Ε, στις μεταφορές ε, έχουμε να κάνουμε με επίγειες μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές. διαλειτουργικότητα, πολυτροπικότητα των ειδών μεταφορών, η η ενέργεια παίζει και αυτή πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λόγω των μετασχηματισμών στις αγοράς ενέργειας. Ε, αναζητούνται πηγές ενέργειας ανανεώσιμες, καθαρές και τα δίκτυα έτσι κι αλλιώς ενέργειας γίνονται ολοένα και πιο αποκεντρωμένα. Ε, η ψηφιακή οικονομία αναφέρεται όχι μόνο σε ψηφιακές υποδομές αλλά και στις πολιτικές που στηρίζουν τις επιδόσεις αυτές, ψηφιακά δικαιώματα, φάσματα κτλ. Και τέλος υπάρχει το θέμα των ανθρώπων, της επικοινωνίας ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα. Ενισχύουμε λοιπόν την συνδετιμότητα ανάμεσα στους πληθυσμούς των δύο περιοχών, στον τομέα της, του πολιτισμού, της υγείας κτλ. Τώρα, εμείς εργαζόμαστε σε διμερή κυρίως βάση με τους δικαιούχους, αν θέλετε, των υποδομών σε συνεργασία με χώρες οι οποίες έχουν δικές τους πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας όπως η Κίνα αλλά και άλλες χώρες οι οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα. Υπάρχει περιφερειακά, υπάρχουν περιφερειακά χαρακτηριστικά σε αυτά τα οποία κάνουμε. Υπάρχουν προγράμματα και δράσεις που διαπερνούν τις μεθορίους και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με περιφερειακά όργανα όπως το ΑΣΕΑΝ και άλλα και αντίστοιχα στην Κεντρική Ασία. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με διεθνείς οργανώσεις επίσης στενότερα γιατί είναι από τους βασικούς αν θέλετε εταίρους που καθιστούν τα δίκτυα διαλειτουργικά και αποτελεσματικά. Και τέλος υπάρχει το θέμα των επενδύσεων στα πλαίσια του επομένου ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τα μέσα τα οποία απαιτούνται εγγυήσεις ε, στον τομέα των, της εξωτερικής δράσης προβλέπονται 60 δις μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν επίσης στον τομέα των δημοσιονομικών ή μάλλον στον τομέα των χρηματοπιστωτικό ε, αρκετοί συνεργάτες όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Δέλτα Νιτάφ και η, τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, ανοικοδόμησης και υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, στους οποίους προσπαθούμε να παρέμβουμε θέματα ανταγωνισμού, θέματα χρηματοδότησης που αφορούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Έχουμε να κάνουμε με τράπεζες που δεν λειτουργούν πάντα σε επίπεδο εμπορικού κινδύνου ε, και επίσης με πιστοτικά ιδρύματα που προέρχονται από άλλες χώρες τα οποία έχουν κρατικές εγγυήσεις όπως η Κίνα. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική θα έλεγα ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες στρατηγική για την δημιουργία των δικτύων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Παρέχουμε λοιπόν ένα σαφές οικονομικό πλαίσιο, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή στην παρούσα φάση. Θα συνεργαστούμε φυσικά με, τις, με, τα, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις μεμονωμένες χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαφής η παρουσίασή σας. Νομίζω ότι ανοίγει τη συζήτηση και για τα θέματα ευρύτερης πολιτικής. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα. Τρεις ερωτήσεις πρώτα και μετά θα ζητήσω από τους ομιλητές. Θα ζητήσω όμως από τους ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις και να μην κάνουν απλές πολιτικές δηλώσεις γιατί αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συζήτηση που θα ακολουθήσει. Έχω τρεις ερωτήσεις. Τι συνδέει την ευρωπαϊκή αντίληψη και την κινέζικη αντίληψη. Ανταγωνισμός, συνεργασία, τι κάνουμε. Δεύτερον, Έχουμε μια ενιαία άποψη σαν Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην κοινωνική στρατηγική. Ε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τις προτιμήσεις των μεμονωμένων χωρών. Ποιος ωφελείται, εν πάση περιπτώσει, από την πρωτοβουλία την κινέζικη. Ακούω ότι συνοδεύεται η πρωτοβουλία αυτή με πάρα πολύ υψηλές δανειοδοτήσεις προς πολλές χώρες. που δεν είναι σε θέση από μόνες τους να ενισχύσουν την οικονομία τους και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται μια κάποια μορφή εξάρτησης από την κινέζικη χρηματοδότηση. Ποιος ωφελείται λοιπόν πραγματικά από αυτού του είδους τις ενέργειες. Μια ερώτηση από τον κύριο Σόλτς. Σας ευχαριστώ για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις σας. τέθηκε ήδη το ερώτημα του Προέδρου. Ποιος ωφελείται και ποιος είναι ο ηγέτης. Ο ηγέτης φυσικά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Αυτή είναι η γεωπολιτική αντίληψη την οποία έχει. Συμφωνούμε λοιπόν ότι η γεωπολιτική και η γεωοικονομική α, αντίληψη είναι συμβατές. Και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά ποιοι είμαστε εμείς από την άλλη που αντιμετωπίζουμε τις συμφωνίες αυτές και τα προγράμματα αυτά. Είναι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ποιοι λοιπόν από ευρωπαϊκή πλευρά, από την ευρωπαϊκή πλευρά είναι σε θέση να χαρακτηριστούν ως συμμετέχοντες στην συμφωνία ή μάλλον στην προοπτική που ανοίγουν οι Κινέζοι. Για τα γεωοικονομικά επαναλαμβάνει ο μιλητής. είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε την αηφορία στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών οι οποίες συμμετέχουν. Κεντρική Ασία ας πούμε. Μήπως εμείς ως Ευρωπαίοι μπορούμε να προτείνουμε κάποιες διαφορετικές απαντήσεις από αυτές τις οποίες θα κατέλεγαν από μόνοι τους εύκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για όσα μας εξήγησαν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για μας συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Δεν έχω καταλάβει. Αυτή όλη η πρωτοβουλία τι, από τι είδους διαχείριση διαπαιτεί, τι γίνεται, πώς γίνεται η επιλογή των έργων, η σχεδιασμός αυτών, ποιος ε, διαλέγει του τους δικαιούχους επιχειρήσεις, πώς είναι δυνατόν να έχουμε κάποιες εγγυήσεις ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα το κάνουν αυτό επίσης ώρες, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Άλλη ερώτηση. Έχουμε κάποια αξιολόγηση των επιπτώσεων όσον αφορά τους στόχους που επιδιώκονται από αυτήν την πρωτοβουλία. Δηλαδή, απασχόληση, κλίμα, ενανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερη συνδεσιμότητα. Έχουν όλα αυτά ζυγιστεί. Άλλο. Θα έχουμε κάποιο είδους παρέκκληση Πρόκειται να γίνει μια μετακίνηση των ε, μεταφορικών ροών από τη θάλασσα προς την ξηρά στο μέλλον. Δεν είπατε τι θα γίνει σε επίπεδο εμπορίου. Τι προοπτικές υπάρχουν. Τι επιπτώσει θα έχει αυτή η πρωτοβουλία όσον αφορά τι ε, εμπορικέ σχέσει ε, Ευρώπη-Κίνα. Thank you. And uh, another question from uh, Salvatore Chiku, and then we'll move to uh, answer κύριος Τσίκου. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Έτσι μπορέσαμε να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας από την ποιότητα των είπανε, από τις ικανότητές τους κλπ. Ακριβώς. Θα ρωτήσω το ίδιο με τους συναδέλφους. Θα ήθελα να μάθω. Πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες ε, διασυνδεσιμότητας σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή. Τι γίνεται με τις ε, κρατικές προμήθειες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τους Ευρωπαίους. Ή θεωρούν οι μας ότι υπάρχουν ε, κάποιοι κίνδυνοι γεωπολιτικοί όσον αφορά την επέκταση των Κινέζων προς την Ευρώπη ή το αντίστροφο. Έχουμε πλέον εκτήματα, έχουμε μόνο κινδύνους. Και τι προτείνουν οι ομιλητές. Τι να κάνουμε. Στην καρδιά του Δήματος παραμένει το πώς δύο τόσο διαφορετικές οικονομίες μπορούν να συνεργαστούν όσον αφορά αυτή την διασύνδεσιμότητα. ρυθμιστικά, κοινωνικά κλπ. Απέχουμε πάρα πολύ. Για να. Πάρα πολύ μεστές ερωτήσεις που προκαλούν προβληματισμό. Φρανσουά, θέλετε το λόγο. Πολύ σωστά το είπατε, Πρόεδρε. Είναι συνεργασία ή ανταγωνισμός, κύριε Πρόεδρε. ανταγωνισμός είναι. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Κινέζοι για την Κεντρική Ασία, τι κάνουν για την Αφρική εμπορικά. Πολλοί βουλευτές ρώτησαν για τις προμήθειες, για τους κανόνες που διαβούν αυτή την υπόθεση. Τελείως διαφορετικό σκηνικό για τους Κινέζους. το Τρασανατόλια, ο δρόμος του μεταξιού. Μα δεν θέλησαν οι συνήθεις χρηματοδότες να καλύψουν τον αγωγό φυσικό Με τα Βαλκάνια εμείς Έχουμε κάποια σχέδια για το μέλλον, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Εν πάση παραμένει η χαόδη απόσταση μεταξύ ημών και εκείνων. Έντερ. Για να τα πούμε όσο γίνεται συνθετικά. Συνεργασία ή ανταγωνισμός. Και εγώ σας παραπέμπω με τη σειρά μου σε αυτά που είπε η Ελλάδα εξ μου. Έχουμε κάποια προηγούμενα όπου έχουμε κάποιες αναπτυξιακές τράπεζες και, και Ιαπωνέζικες που χρηματοδοτούν τις χώρες που κερδίζουν κάποιες συμβάσεις. Να ο ανταγωνισμός. Φυσικά υπάρχουν και επικαλυπτόμενα συμφέροντα έχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας, αλλά ως εκ το πλήστον. Επειδή το κίνητρο είναι να επεκταθεί η κινέζικη οικονομία για να βοηθούν οι εταιρείε του, ε, βέβαια, πρόκειται περί ανταγωνισμού. Ποιο ωφελείται, ήταν άλλη ερώτηση. Αν πλευρά Κινέζων υπάρχουν πολλά ωφέλη αλλά και κίνδυνοι για τι χώρε που φιλοξενούν αυτά τα έργα. Τι γίνεται τώρα από πλευρά Ευρώπης. Είδαμε από πλευρά ε, Κίνας τα πράγματα πριν αλλά τώρα πλευράς Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι τα συμφέροντά μας είναι να έχουμε κάποιους κανόνες, να έχουμε κάποια πρότυπα όπως ο κ. Αυτά δεν τα έχουν αναγκαστικά και οι Κινέζοι όσον αφορά αυτή την υπόθεση. σε σχέση με το αν υπάρχουν πάντα διαγωνισμοί, αν υπάρχει χρηματοδότηση από κάποια μεγάλη κρατική τράπεζα. Έχουμε τις εξαγωγικές ε, ε, εγγυήσεις, τις κρατικές, τις κινέζικες. Για το BRI. Έχουμε απαντήσεις. Στα Βαλκάνια που είναι τόσο κοντά στην Ευρώπη, Εκεί να έχουμε κάποια απάντηση. Έχουμε το να έχουμε προσχώρηση αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε πιο γρήγορες διαδικασίες συνεργασίας. Τώρα ποιος ελέγχει τον BRI. Δεν υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων ενιαία. Το πράγμα είναι σπασμένο στις κοινωνικές επαρχίες, στα διάφορα υπουργεία. Πρέπει να εξετάσουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Ε, τα είπε και ο συνέλφος από την πρεσβεία και θα πρέπει να εξετάσουμε ποια έργα κατατείνουν στην επίτευξη των στόχων. υποδομές, ψηφιακή τεχνολογία και οι εμπορικές ροές. Τώρα, πριν ολοκληρώσω, είναι κάτι που δεν το αναφέραμε τόσο πολύ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι στρατηγική που έχει η Κίνα που και την έχει πολύ πριν αυτή την πρωτοβουλία, αλλά τώρα έχουν εντείνει τις προσπαθίες τους. Το βλέπουμε στις ομιλίες ηγετών, διάφορες ομάδες εργασίας, έχουν συγκεκριμένα αποτέλεσματα αποσπάσει με την Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου, με την Γεωργία, Μολδαβία. Θα προχωρήσουν με αυτή τη στρατηγική, ιδίως σε χώρες που έχουν DCFTAs, ανοψιακές ε, συμφωνίες με την Ευρώπη. Και έτσι η Κίνα μέσω ε, αυτών των τρόπων, οι πλατφόρμες που λέμε, θα μπει στην Ευρώπη, ούτως Γεια, Η Άστρεντ, πολλά ακούσαμε. Δεν θα ξεκινήσω λοιπόν να αναφέρουμε σε κάθε από από τα στοιχεία αυτά. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για το θέμα της συνεργασίας και του ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Θα πρέπει να εξετάσουμε ότι είναι πολλές οι χώρες που συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία αυτή. Δεν είναι λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο με την Κίνα γιατί έχει να κάνει με τις χώρες αυτές. Ε, αν κοιτάξουμε τι γίνεται στην Κεντρική Ασία, για παράδειγμα, έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες χώρες. Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν αναφέρθηκε στη, Ρωσική, στη Ρωσία και στην ε, Ρωσική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά την ε, Ασία, στο Καζακστάν. Πολλά ακούσαμε, αλλά δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε συζητήσει συγκεκριμένα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οι αλλαγές και εξελίξεις στο Καζακστάν και αλλάζει ακόμα Πιστεύω ότι αυτό ε, ενδιαφέρει και την ευρωπαϊκή διάσταση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το διμερέ επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, αλλά και σε ό,τι αφορά την συνολική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κεντρική Ασία. Δεύτερο θέμα. Επειδή συζητήθηκε τα θέματα διακυβέρνηση, κατά πόσον υπάρχει μια πλατφόρμα και κατά πόσον λειτουργεί και πώ. Το είπα και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει κάποια σαφής χώρια διαχείριση για το θέμα αυτό στην Κίνα. Υπάρχει μια πληθώρα διαδικασιών. Για μας λοιπόν αυτό είναι πολύ ασαφές ως σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης. Πάντα θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. και περνάμε το ποτάμι ακουμπώντας τις πέτρες στο πυθμένο του ποταμιού. Είναι πολύ κινέζικη αυτή η προσέγγιση. Δεν υπάρχει λοιπόν μια διεθνής πλατφόρμα που μπορεί κανείς ε, να εξετάσει όλα αυτά τα project. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα και για την ε, φυσική ε, συνδεσιμότητα και για τη θεσμική συνδεσιμότητα. Και σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα μεταξύ ανθρώπων. Πολλά ακούσαμε για το soft power και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την ε, Κεντρική Ασία. Δεν υπάρχει λοιπόν μια κεντρική πλατφόρμα για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έχουμε τέσσερα λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Και έχουμε και δύο άτομα τα οποία ενδεχομένω να θέλουν να πάρουν το λόγο. Να προσπαθήσουμε να σας ακούσουμε και τους δύο, μάλιστα. Τηλεγραμματικά. Επιγραμματικά, συγγνώμη. Καταρχάς, η στρατηγική αυτή είναι η ενσωμάτωση της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της εμπειρίας που έχουμε και με την ενιαία αγορά για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόκειται για πρότυπα περιβαλλοντικής ε, προστασίας ε, βάσει των βελτιστών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και νομίζω ότι αυτό θα καταστεί όλο και πιο ε, ελκυστικό για χώρες όσο ανεβαίνει το επίπεδο τους. Κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του BRI αναφέρεται την σχετική πλατφόρμα συνδεσιμότητας η οποία είναι υπό επέκταση. Κοιτάμε τώρα τη συνεργασία σε τρίτε χώρες στο πλαίσιο τη στρατηγική μα και του BRI. Κατά πόσον υπάρχει μία προσέγγιση στα κράτη-μέλη. Όντω υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη στρατηγική μα που τα πετύχαμε και υπήρχε μεγάλο επίπεδο σύγκληση σε ό,τι αφορά ακριβώ το μοντέλο το οποίο έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο είναι το ευκταίο όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Τίθεται επίση το θέμα του ποιο ωφελείται από τα προγράμματα αυτά. Είναι δύσκολο να αποφανθούμε γιατί δεν έχουμε διαφάνεια. Το ξέρουμε ότι το BRI πάει πιο καλά σε χώρες ε, με λιγότερη καλή διακυβέρνηση από τις χώρες με καλή διακυβέρνηση. Επίσης σημειώνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά το ποσοστό χρέωσης, κάποια από τα παραδείγματα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το Πακιστάν σήμερα πιστεύουμε ότι κάπως θα πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τις άλλες χώρες Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία. Θα έχει και τον παράγοντα συνδεσιμότητας αυτή η στρατηγική. Και στο σημείο αυτό θα βάλω τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο. Ευχαριστώ και θα είμαι σύντομο. Νομίζω ότι συμφωνούμε ουσιαστικά σε ένα σημείο ότι η πρωτοβουλία BRI δεν είναι η μοναδική προτεραιότητα που θα μπορούσε να επιφέρει ευημερία σε όλη την Ήπειρο και συνδεσιμότητα. Είναι μόνο μία από τις προτεραιότητες αυτές και μία από τις ε, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Ξεκίνησε από την Κίνα. Δεν είναι μόνο της Κίνας, έχει διπλάσιο πολλαπλασιαστό και θα επιφέρει ε, ε, αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Έννοιας και της στρατηγικής συνδεσιμότητας. Εγώ πιστεύω ότι σαφώ επικρατεί η συμπληρωματικότητα και όχι τόσο πολύ ανταγωνισμό. Και να είμαι ειλικρινή, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς συνεργασία. Και είναι γεγονό ότι έχουν ξεκινήσει Συζητήσει σε ό,τι αφορά τι πλατφόρμες ε, συνδεσιμότητας. Και τρίτον, ποιο θα ωφεληθεί. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολλά ωφέλη και για την Κίνα, θα ωφεληθεί ασφαλώς και κάποιες χώρες επίσης θα ωφεληθούν. Η Siemens της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχει συνεργαστεί με πάνω από 100 ε, για να φτιάξει γεννητρίες για αφρικανικές χώρες. Μέχρι τα τέλη του 2020 θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Η Car Express έχει ε, αυξήσει κατά 10.000 ε, τις πωλήσει. Το Αμβούργο περίπου 600 ε, γερμανικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις μας. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και λάβαμε πολλές απαντήσεις. Κάποια από τα ζητήματα παραμένουν εκκρεμή, ενδεχομένως να απαντηθούν δεύτερη, ε, στο δεύτερο πάνελ. Έχουμε ένα πάνελ με τέσσερα μόνο άτομα. Το ερώτημα είναι πώς θα τεθεί στην πρακτική το θέμα η συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Πρώτος ομιλητής, Μάγια Μπάκραν Μάτσιτς. Ελπίζω σωστά να, να προφέρω το όνομά σας, η οποία είναι και γενικός γραμματέας για... Συγγνώμη, ε, Διευθύντρια, Γενική Διευθύντρια για την Κινητικότητα και στη Μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Τομπία δεν έχει από τη Siemens. Η γερμανική εταιρεία υποδομών, ο κ. Φραντσέσκο Ρώση, ο οποίο είναι ιδρυτή τη TechSeal και θα μα εξηγήσετε εσεί τι κάνετε ακριβώ στον τομέα των ψηφιακών για τα θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Και ο κ. Τιμ Ντεμάιερ, ο οποίο είναι υψηλό βαθμό σύμβουλο του ΠΟΕ. Θα μα μιλήσει για την πλευρά της απασχόλησης του θέματος της συνδεσιμότητας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν ε, είμαστε ακόμα πολύ οριακά, χρονικά, αλλά παρακαλώ όχι παραπάνω από 5 έως 7 λεπτά για να έχουμε περιθώριο να συζητήσουμε μετά. Yeah. Thank you. Mm. Thank you very much and... Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω με τη χαρά συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση και να ευχαριστήσω τους ομιλητές στο πρώτο πάνελ και να πω όταν μιλήσατε ε, για, την, για τον ανταγωνισμό ε, και τη συνεργασία αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι παρά τον ανταγωνισμό απαιτείται η συνεργασία Τώρα, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στον τομέα των μεταφορών, πάρα πολύ σύντομα, θα παραπέμψω σε αυτό που ονομάζουμε, σε αυτό που ορίζουμε εμείς σαν συνδεσιμότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Υπάρχουν τρία στοιχεία. Καταρχάς, εμπειρίες στον τομέα της δημιουργίας δικτύων για να δημιουργηθούν διαμεθοριακές συνεργασίας, Εταιρικέ σχέσεις ε, με χώρες και λαούς και τρίτον ε, βιώσιμη χρηματοδότηση. Τώρα για τη δημιουργία συνδέσεων και τις εταιρικές σχέσεις. Τι εμπειρίες μπορούμε εμείς να μοιραστούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπετε ε, τα TENS. Έχουμε κάνει δεκτά τα πρώτα προγράμματα ήδη από τη δεκαετία του 90 και είναι βασικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής αγοράς. Τα τέντι βασίζονται στην εφαρμογή κανόνων και αρχών, κανόνων και αρχών που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου. Τα TNT λοιπόν έχουν υιοθετήσει την δικτυακή αντίληψη εμείς δίδουμε συγκεκριμένη προτεραιότητα σε προγράμματα κοινού συμφέροντος ε, στα πλαίσια της συνοχής και της διαλειτουργικότητας των TENS. Με άλλα λόγια, το ten είναι μία σειρά ε, δικτύων μεταφοράς ε, επίγειας, θαλάσσιας, εναέριας τμήμα ενός συστήματος που περιλαμβάνει επίσης δίκτυα ενέργειας και δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις οδικές μεταφορές, τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις αερολιμενικές εγκαταστάσεις, την κατασκευή ε, οδών υψηλής ταχύτητας και έχουμε επίσης ε, και τα ίδια επίπεδα και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ασφάλειας. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να περνάει από μια εξαντλητική ανάλυση ωφέλους και κόστους, χρηματοδοτική ανάλυση, όπως επίσης και η φόρο ανα, ανάπτυξη, κάτι το οποίο ε, επηρεάζει φυσικά το θέμα του περιβάλλοντος. Και φυσικά θα πρέπει να ωφελούνται όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε αποκτήσει πολλές εμπειρίες τα τελευταία 20 χρόνια. Όταν βλέπουμε το πώς αναπτύσσονται τα δίκτυα σήμερα, βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα είναι σχετικά επιτυχή και δίδουν αποτελέσματα. Με λίγα λόγια αυτά είναι τα στοιχεία εμπειρίας τα οποία μπορούμε να μοιραστούμε με τους εταίρους μας στην Ασία. Και σε αυτά θα αναφερόμαστε όταν ξεκινήσουμε και από κοινού κάποια προγράμματα. Τέτοια προγράμματα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να αποδώσουν εφόσον υπάρχουν σωστές διαβουλεύσεις με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των ΤΕΝΤΗ είναι οι διαμεθοριακές συνδέσεις και εδώ έχουμε σημαντικές εμπειρίες αποκτήσει. Είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα των ΤΕΝΤΗ, οι διασυνοριακές συνδέσεις και αυτό μας έχει επιτρέψει να συνδέσουμε σωστά το βορρά με τον νότο και την ανατολή με τη δύση. Ήδη έχουμε μια νομικά δεσμευτική διεύρυνση των TNT και στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες ε, ε, της, Δυτικής, ε, της Κεντρικής Ασίας και γενικότερα στις χώρες της Μεσογειακής Δεκάνης. Η Συμφωνία Διεύρυνσης των Δικτύων ελήφθη από κοινού με τους εταίρους Έρχομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας μου για το πώς συνεργαζόμεθα με την Κίνα, εφόσον συνεργαζόμεθα με την Κίνα. Έχουμε δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε πλατφόρμα συνδετικότητας και αναφέρθηκαν σε αυτήν πολλοί ομιλητές πριν από μένα. Η πλατφόρμα αυτή είναι στην ουσία ένα βήμα για διάλογο. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στη στρατηγική της Κίνας και την πολιτική μας στον τομέα των στρατηγικών υποδομών. Στις διαφάνειες αυτής βλέπετε τις διαφορετικές μορφές σύνδεσης ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως εδώ έχουμε σταθεί περισσότερο στις επίγειες συνδέσεις. Στην τρίτη πλατφόρμα που έγινε στο Πεκίνο τον Ιούλιο προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή έρευνα για τις πιο βιώσιμες ιοδρομικές συνδέσεις ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη. Έδειξε ε, τη δυναμική ορισμένων συνδέσεων και τις πιο ρεαλιστικές συνδέσεις, του πιο ρεαλιστικούς και αποδοτικούς διαδρόμους. Είδαμε ότι αυξάνονται συνεχώς οι σιωδρομικές μεταφορές και γι' αυτό είπαμε με τους εταίρους μας στην Κίνα ότι και με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας θα εξετάσουμε τους σιδηροδρομικούς αυτούς διαδρόμους και να δούμε τι είδους υποδομές απαιτούνται περαιτέρω. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να εντοπιστούν οι πιο αποδοτικοί ε, σιδηροδρομικοί διάδρομοι. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις ε, ισχύουσες συνθήκες σήμερα και τις εμπορικές ροές. Έχουμε σαν στόχο να βελτιστοποιήσουμε τις συνέργειες ανάμεσα στα τέντη και τη στρατηγική των Κινέζων. Αυτό κάνουμε λοιπόν σε συνεργασία με την Κίνα, με επικοδομητικό τρόπο νομίζω και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί τους τις εμπειρίες τις οποίες έχουν συλλέξει εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλές φορές γράφουμε στα προγράμματά μας ε, ότι οι, τα τεντή συναντούν την κινέζικη στρατηγική. Επόμενος, ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνει την ευκαιρία να σας πούμε την γνώμη μας όσον αφορά αυτήν την ε, πρωτοβουλία από δική μας πλευράς να είμαι σύντομος Τρία θέματα θα σας πω. Να συμπληρώσω για αυτά που ακούστηκαν. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ευρύτερη οπτική ε, όσον αφορά την διασυνδεσιμότητα γιατί δεν πρόκειται μόνο για μεταφορές είναι η σύνδεση της μίας χώρας με την άλλη με σιδηρόδρομο, δρόμους, λιμάνια, άρα εδώ μιλούμε για πολύ περισσότερα πράγματα. Να, ποια θα πρέπει να είναι η στατική. Καλύπτεται και η ηλεκτρική ενέργεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι η βασική υποδομή είναι επίσης και η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Γι' αυτό και φτιάχνουν τώρα τον δρόμο του μεταξύ των ψηφιακό. Άρα, για να δούμε. Κάτι που θεωρούμε ότι επίσης μας δίνει περισσότερες δυνατότητες σε εμάς και στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Άρα, δεν μιλάμε μόνο για την ε, υλική συνδεσιμότητα. Είπαμε να διευρύνουμε το φάσμα αυτής της πρωτοβουλίας. Το BRI, να δούμε τι ωφέλη μπορεί να προκύψουν, τι θα γίνει με το Belt and Road και υπήρχε και μια πρόδρομη φάση πριν αρχίσει το ίδιο το Belt and Road Δηλαδή είχαμε κάποια υποστήριξη, χρηματοδοτική, ε, συνέβαιναν πράγματα πολύ πριν το 2013. Στη Γερμανία είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι, έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας σε σχέση με την επιχειρησιακή μας, επιχειρηματική μας επιτροπή. Προσπαθούμε να καλύψουμε εταιρείε, προσπαθούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το Belt and Road για να μπορούμε να δούμε τι κοινέ ευκαιρίες υπάρχουν. Να μην ανταγωνιστούμε τους Κινέζους αναγκαστικά, να συνεργαστούμε. Για μας είναι ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα στρατηγικής ε, Ευρώπης-Ασίας. Είναι κάτι το παγκόσμιο, ξεκαθαρίστηκε από τους ομιλητές. Αφορά και τις Ομένες Πολιτείες, Ινδία, Ιαπωνία επίσης. Και ήδη έχουν εμπλακεί δεν είναι απειλή, είναι δυνατότητες για όποιες εταιρείε θέλουν δυναμικά να δουν τι, τι, προσφέρεται. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όχι μόνο με την Κίνα αλλά για όλες τις σχολές του BRI. Όλοι όσοι λαμβάνουν κάποια ενίσχυση για αυτή την υποδομή, αυτές τις υποδομές. αν έχουμε σοβαρές προθέσεις ε, θα πρέπει σε συνεργασία και με τους άλλους Αμερικανούς και Κινέζους να καταλάβουμε τις ανάγκες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και έτσι να αντιδράσουμε, να ανταποκριθούμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε ως Ευρωπαίοι, ως Γερμανοί, το ίδιο κάνει και η Ζημενς. Είναι ευκαιρία να δούμε πως κάποια έργα δεν είναι βιώσιμα, δεν χρειάζονται πραγματικά να συνεργαστούμε, να καταλήξουμε σε κάτι το βιώσιμο. Όπως είπαμε. Τώρα είναι κατάλληλη στιγμή γιατί μετά από πέντε χρόνια θεωρούμε το, το BRI είναι σε μια καλή φάση και μετά τον αρχικό ενθουσιασμό μετά από κάποιες ε, επικρίσεις βλέπουμε ότι κάποιες χώρες τελικά δεν εγκαταλείπουν, ε, εξετάζουν τα πράγματα. Υπάρχει θετική τάση. Το BRI δεν έχει φρενάρει, απλώς μπορεί να αλλάξει μορφή. Προσοχή, μήπως τελικά έχουμε ένα βάγιο δημοσίων σχέσεων για το θέμα. Άρα τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο πολύ, οπότε κάνουν το Belt and Road δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Μιλούμε περισσότερο στη Γερμανία και στην Ευρώπη για συνεργασία. Μεγάλη ευκαιρία. Να την αδράξουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε. Βοήθεια προς την Κίνα, βοήθεια και στις χώρες που θα υπάρξουν υποδομές. Να, αυτά πρεσβεύει η Siemens σχετικά. Εδώ και πολύ καιρό η Κίνα είναι τέρο όλων αυτών των χωρών. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να προσθέσουμε άλλη μια διάσταση. Τη διάσταση προσυδειάζει στη διάθε χώρα. ένα σωρό χώρες. Βοηθούνται από την Ρωσία. Εργαστήρια, διερεύνηση του πραγματικά χρειάζεται και άρα να δούμε τι δυνατότητες έχουν οι Κινέζοι. Μετά να πάμε στην Κίνα για να βρούμε συνομιλητές. Ναι, σας θέλουμε, λέμε, για εταίρο αλλά η Siemens θέλει να υπάρξει δημιουργία θέσεων εργασία, χρειαζόμαστε διεθνή πρότυπα. Ε, αυτά θα υπαγορεύσει η Siemens. Και μετά να δούμε τι λύσεις υπάρχουν για το έργο. Και οι Κινέζοι γιατί όχι μπορεί να εντυπωσιαστούν από τις ιδέες που τους προσφέρουν και δεν έχουν. Οπότε λοιπόν δεν έχει να χτυπήσει την πόρτα, θα πρέπει να ψάξουν οι εταιρείε οι γερμανικές να δουν ε, δυναμικά, να αποταθούν στου Κινέζους, να δουν και να μάθουν τι συμβαίνει. Α, και τελευταίο. Πολύ καλό να έχουμε το Made in Germany. Όμως, το Made in Europe θα πρέπει να είναι κάτι που να, πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο καμία χώρα δεν μπορεί να καταφέρει μόνη τη. Η Ευρώπη όλοι μαζί. Άρα αυτή η στρατηγική connectivity για την συνδεση μόντα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και να μην πάμε μόνο προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού. Να δούμε πώς θα λύσουμε τα σύγχρονα προβλήματα με συνεργασία μέσω αυτών των έργων. Το Μπάιας, ευχαριστούμε να σας... εξηγήσω αυτά τα οποία κάνουμε μέχρι τώρα. Καταρχάς εμείς ε, φέρνουμε σε επαφή τις νεοφυείς επιχειρήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με επενδυτές από την Κίνα και βοηθούμε έτσι στην ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες υπάρχουν στη μία ή στην άλλη πλευρά κάτι το οποίο ε, γίνεται κυρίως από πλευράς ε, ε, όπως είπα Κινέζων επενδυτών οι οποίοι όμως δεν ελέγχουν τις διαδικασίες στον τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη και όλα ελέγχονται από πλευράς Ευρωπαίων διαχειριστών. θα μπορούσα να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα το τι σημαίνει για μας η κινέζικη στρατηγική. Αναφερθήκατε στη συνεργασία, αναφερθήκατε στον ανταγωνισμό και στην ψηφιακή συνεργασία. Η νέα πρωτοβουλία των Κινέζων, το BRI, δεν είναι ξεκάθαρο αν καλύπτει και ποιους τομείς. Δεν ξέρουμε αν περιορίζεται στις μεταφορές Ο πραγματικός ανταγωνισμός μέχρι τώρα ε, που αφορά στη Γερμανία ή και το σύνολο της Ευρώπης δεν είναι η Κίνα που ανταγωνίζεται την Ευρώπη αλλά με μονομένες ε, περιοχές της Ευρώπης ε, που ανταγωνίζονται η μία την άλλη στην Κίνα μέσω των γραφείων του. πριν γίνει μια κοινή πρόταση απαιτούνται πάρα πολλές συναντήσεις έτσι ώστε να υπάρξει ο ελάχιστος επιθυμητός συντονισμός. Καταρχάς θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Κίνα έχει αλλάξει. Η άποψη είναι ότι η Κίνα στην ουσία κατασκευάζει πράγματα. Αλλά ξεχνάμε ότι η Κίνα ταυτόχρονα καινοτομεί και αναζητεί τεχνολογία για να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και στην ίδια της την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ακόμα δηλαδή η Κίνα στον τομέα της έρευνας όχι τόσο για τις εξαγωγές, αλλά για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν οι κοινοζικές επιχειρήσεις ε, στον εσωτερικό της χώρας. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ σημαντικά, 1,63 στην ε, ψηφιακή οικονομία στην Κίνα. Ε, είναι μια αγορά πολύ, πολύ ακριβή να έχει κανείς πρόσβαση βέβαια τι είδους συνδεσιμότητα προβλέπουμε λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχάς θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες να έχουν μια ευέλικτη σχέση ε, η οποία ε, θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν χωρίς ε, να διαρρήξουν τους δεσμούς τους με τις παραδοσιακές τους αγορές. Ταυτόχρονα ο δρόμος αυτός είναι η επικοινωνία με την Κίνα δηλαδή είναι διπλής κατεύθυνσης. Νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να επενδύουμε, να αγοράζουμε μετοχές σε κινέζικα προϊόντα και να επενδύουμε επίσης και σε μικτές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές και κινέζικες έτσι ώστε να σταθμίσουμε κάπως καλύτερα τους κινδύνους. Κάνοντας το αυτό, στην ουσία δίδουμε υψηλές πιστώσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κίνα και υπάρχουν ταυτόχρονα πάρα πολλές ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται σε επίπεδο του προϋπολογισμού τους από μεμονωμένους Κινέζους επενδυτές. Το θέμα είναι να υπάρξει μια σωστή μορφή συνεργασία και όχι μόνο ακολουθώντας το, αυτά τα οποία προβλέπει το σύστημα να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλο. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο να μπορέσει με ευέλικτο τρόπο να επενδύσει στην Κίνα χρησιμοποιώντας τις διαθεσιμότητες τις οποίες παρουσιάζει η χώρα αυτή και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τις κοινοζικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν μαζί μας. Γιατί πολλές φορές υπάρχει πάντα μία κάποια απομόνωση. Ο καλύτερος τρόπος είναι να είναι κανείς παρόν στο Πεκίνο. Παρά τους περιορισμούς εμείς έχουμε ένα γραφείο μόνιμο στο Πεκίνο και έτσι κατανοούμε ακριβώς το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναπτύξουμε μια ενιαία αντίληψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, από την Ευρώπη προς την Κίνα και τις μικρομεσαίες γενικότερα στην Κίνα και έτσι θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι το τι μπορούμε να κάνουν για να ενισχύσουν την αγορά αυτή και όχι μόνο να υπόκεινται ε, στις συνθήκες της αγοράς. Η Ευρώπη λοιπόν σε σχέση με τις μικρομεσαίες είναι διαθέσιμη στην Κίνα. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην κινέζικη αγορά. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα συντονισμός των μηχανισμών που βρίσκονται στην Κίνα έτσι ώστε να διευκολυνθούν ακόμα καλύτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην συγκεκριμένη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τώρα να περάσουμε στον Τιμ να περάσουμε από τον κόσμο των ε, εργοδοτών που πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα ήθελα στους εργαζόμενους που ε, πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ποια είναι η άποψή σας από πλευρά του της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που καλέσατε την ε, Δεθνή Οργάνωση Εργασίας εδώ στο πάνελ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις ε, για την εμπορική πολιτική σε ό,τι αφορά και την Ευρώπη, την Ασία και τον παράγοντα συνδεσιμότητα ε, ευρέως. Δεν θα επικεντρωθώ ιδιαίτερα στην Κίνα. Καταρχάς, να πω ότι με σαφήνεια για μας ε, τα τα, οι συνθήκες εργασίας και ε, οι προδιαγραφές εργασίας αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα ε, για το εμπόριο. Αυτό αναγνωρίζεται στην Ευρώπη πλέον και όλο και πιο πολύ στην Ασία. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πάντα ήταν αυτό μια, αν θέλετε, οργανωμένη συνεργασία και τόσο πολύ ένα παθιασμένο, α, μια παθιασμένη συνύπαρξη. Οι εργοδότες με ένα όραμα πριν από 200 χρόνια ήδη είχαν το θέμα ότι ήθελαν να συνεχίσουν ε, να κάνουν ε, δουλειές ε, και να ασκούν το επάγγελμά τους, αλλά να προσφέρουν και σωστούς ε, όρους εργασίας, γιατί και αυτό θα τους απέφερε καρπούς μακροπρόθεσμα. Με έναν τρόπο λοιπόν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι οι ανταγωνιστέ μα θα πρέπει λίγο πολύ να είναι στο ίδιο επίπεδο, να κάνουν λίγο πολύ τα ίδια. Αυτό το λίγο πολύ είναι σημαντικό. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Και αυτή είναι και η επίσημη τοποθέτηση της παγκόσμιου Οργάνωση εργασία, ότι ουσιαστικά αναγνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν νόμιμο συμφέρον στην πολιτική του, στην εμπορική πολιτική του, να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει ένα λίγο πολύ ίσο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη πρότυπα, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερω την εφαρμογή του εργατικού δικαίου και ότι υπάρχει ένα συμφέρον να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες δεν χρησιμοποιούν χαμηλότερες συνθήκες εργασίας ως ε, πλεονέκτημα ιδιαίτερα τέτοιες ε, συνθήκες εργασίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τεχνικές προδιαγραφές. Στον τομέα λοιπόν αυτό δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε μια θέση που να μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει πραγματικά ίση όρια ανταγωνισμού. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία και θα πρέπει να κάνουν τις δικές τους προσαρμογές στο πλαίσιο της σταδιακής έκθεσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Άρα εδώ πέρα ακολουθούμε την αρχή των προτύπων που έχουν τεθεί σε επίπεδο τριμερές για να εξασφαλίσουμε ότι η επικύρωση των τεχνικών προδιαγραφών θα παραμείνει σε θελούσιο επίπεδο. Είναι σημαντική παράλληλα όμως η επικύρωση, γιατί πιστεύουμε παράλληλα ότι τα επιτέχματα τα οποία έχουμε πετύχει δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε να υπαναχωρήσουν. Στο σημείο λοιπόν αυτό στις τελευταίες συμφωνίες ε, απελευθέρωσης που είδαμε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλα τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια. Και από πλευράς διασύνδεσης θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλός τρόπος ε, για να προχωρήσουμε. Η εμπορική πολιτική δεν έχει να κάνει τόσο πολύ μόνο με αριθμητικά στοιχεία, αλλά με μακροπρόθεσμα πλέον εκτήματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, όπως αποκαλείται συχνά σήμερα. Και κάποιες σκέψεις τώρα, αναπόφευκτα, για το πού βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η Ευρώπη σε σχέση με την Ασία. Η Ευρώπη και οι αναπτυγμένες μάλλον χώρες στην ΕΟΣΑ έχουν ε, επικυρώσει 65 συμβάσεις. Στην Ασία είναι πολύ πιο χαμηλό το πόσο αυτό. Κατά μέσο όρο 22 τέτοιες συμβάσεις. Άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία είναι πάρα πολύ διαφορετική εντό των ε, ασιατικών χώρων. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Κορία, το Βιετνάμ και τι Φιλιππίνες, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το νομικό σύστημα, των χωρών. Η κατάσταση είναι και πολύ διαφορετική επίση. και βλέπουμε ότι ναι μεν υπάρχει σεβασμό. και έντονο, ενδιαφέρον για τα διεθνή πρότυπα υπάρχει δισταγμό σε ό,τι αφορά τη δέσμευση. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ε, συνθήκες ε, λόγω των ίσων όρων θα αναμέναμε να επικυρώσουν τα πιο πολλά κράτη-μέλη. Δύο τρίτα των επικυρώσεων, των επερχόμενων επικυρώσεων, είναι από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Οι πιο τεχνικές περιοχές βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί πιο πολύ ενδιαφέρον για την ε, υγεία, την κοινωνική ασφάλεια, λιγότερο όμως στο θέμα το μεστολογικός οι επικυρώσεις για την προστασία των μισθών, για τον κατώτατο μισθό, την προστασία μισθού, όταν ε, υπάρχει υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμό κτλ. Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξή: ότι έχουμε εκπροσωπήσεις και διαδικασίες καταγγελιών, αλλά λίγες είναι τελικά οι περιπτώσεις που προωθούνται στην περιοχή και αν τη συγκρίνουμε την κατάσταση με τη Λατινική Αμερική είναι μεγάλη διαφορά. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά πρότυπα υπάρχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο ότι τα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, το επιχείρημα των ανθρωπινών δικαιωμάτων γενικότερα δεν παίζει ιδιαίτερα. Αλλά οι εμπορικέ συμφωνίε καταδεικνύουν ε, συστηματικά ότι έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση των εργασιακών προδιαγραφών και στην πολιτική ατζέντα. Ε, μίλησα πολύ ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μιλώ μόνο για τα θεσμικά όργανα, αλλά και οι εταιρείε ε, που επενδύουν στην Ασία, θεωρώ ότι έχουν πολύ σημαντικό ηγετικό ρόλο να διαδραματίσουν για να εξασφαλίσουν κάποια συνδεσιμότητα η οποία θα είναι πέρα από το επίπεδο το άμεσο οικονομικό, πέρα από τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα και νομίζω ότι η πρόσφατη συνθήκη έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσει, αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση για το Βιετνάμ. Αποτελεί ένα πολύ καλό μοντέλο. Και βάσει τη έρευνα που κάναμε σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα εργασιακά, διαπιστώνουμε ότι τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και οι κοινωνικές αυτές ρήτρες να καταστούν πιο εφαρμόσιμες. Γιατί δεν έχουν συμβεί πολλά από την άποψη αυτή και να μην ξεχνάμε ότι, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ για κάποια από τα εργασιακά αυτά πρότυπα πραγματικά χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, μεγαλύτερη ικανότητα, πρωτοβουλίε ε, σε ό,τι αφορά την επιμέλεια, σε ό,τι αφορά ε, την ε, διαφάνεια των πολυεθνικών εταιριών πολύ σημαντικά ζητήματα. Έχουμε και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι πολυμερεί τράπεζε, όπω η Ασιατική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και να περάσουμε λοιπόν τώρα γρήγορα στι ερωτήσει, λέει η Πρόεδρο. Και πραγματικά έχουμε λιγότερα από 15 λεπτά στη διάθεσή μα για ερωτήσει αυτή τη φορά. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο λοιπόν για να θέσει το πρώτο ερώτημα. Μία πλήρη ερώτηση ο Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και φυσικά αναπτύσσουμε ε, εμπορικά μέτρα, συζητάμε τέτοιες, ε, τέτοια μέτρα. Έχουμε το παραδοσιακό, αν θέλετε, τα παραδοσιακά εργαλεία για το εμπόριο, εμπορικές συμφωνίες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πώς ε, αυτή η εμπορική εργαλειοθήκη μπορεί να ταιριάξει στο ζήτημα της συνδεσιμότητας και είναι περίπλοκο το θέμα αυτό γιατί έχουμε διάφορους διάφορες χώρες, διαφορετικές υποδομές. Ποια θα ήταν λοιπόν η σύσταση για τις περαιτέρω εμπορικές συμφωνίες. Άλλη ερώτηση από το κοινό, ο κύριος Σόλτς. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ενδιαφέρον το ότι μιλήσαμε για την ανάπτυξη τέτοιας εργαλειοθήκης. Αναρωτιέμαι όμως αν είμαστε έτοιμοι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και για παράδειγμα, βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η τάση της ζήμησης της να συνεργαστούν για να, κάνουν, να, δημιουργήσουν πιο ισχυρό ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δραματίσει πιο έντονο ρόλο και να δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πιο πολλές δυνατότητες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ή θα κινηθούμε με 26-27 διαφορετικά εθνικά συμφέροντα και ο καθένα στην τύχη του και μόνος του και μετά θα διερωτώμαστε γιατί δεν συνδεόμαστε. Δεύτερη ερώτηση. Η συζήτηση για την Huawei και το 5G. Τι λέμε για τους Αμερικανούς. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση. η τηλεπικοινωνία στη Γερμανία, για παράδειγμα, και οι εταιρείε είναι προτιμασμένοι να κάνουν τα ίδια που κάνει η Huawei. Τηλεφώνικα τη Ισπανία ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια εταιρεία. Συζητάμε λοιπόν ότι είμαστε σε θέση να συναγωνιστούμε με τις ε, ταχύτατες εξελίξεις ε, στον ψηφιοποιημένο κόσμο, με τις τεχνολογίες. Ή, για παράδειγμα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ίσως ε, θα υπάρχει σαφές πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά το υδρογόνο. Και αφαιρέσουμε τη διάσταση της ηλεκτρονικής οδήγησης, γιατί κανείς δεν ξέρει πού βρισκόμαστε. Δεν βλέπω να υπάρχει προθυμία να υπάρξει συζήτηση προς την κατεύθυνση αυτή, να γίνεται τέτοιο νέο βήμα για τη συμμετοχή στην δραστηριότητα αυτή. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση λέει ο Πρόεδρος. Αν όχι, και κλείνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Θα κάνω και εγώ μία ερώτηση. Μία ερώτηση για τη Μάγια Μπάκραν Μάκριτς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς η γενική σας διεύθυνση, πώς η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, πώς κάνει η σύνδεση με την ε, εμπορική πολιτική, με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συζητήσαμε σε τέτοιες ε, μεταξύ της ε, ατζέντα συνδεσιμότητας. Προφανώς υπάρχει σύνδεση, αλλά πώς γίνεται αυτός ο σύνδεσμος και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η οποία όλο και πιο πολύ συμμετέχει στο εμπορικό αυτό κομμάτι. Θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση εδώ. Και έτσι λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά. Να ναι. ακούσουμε. Να σας πω, να ξεκινήσω Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επηρεάζει όλο και πιο θετικά τις εργασίες μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με όλες τις πλευρές της συνεργασίας με την Κίνα. Και νομίζω ότι από τα στοιχεία τα οποία σας μεταφέραμε μέχρι τώρα έχετε κάποιες απαντήσεις σχετικά με τα εμπορικά μέσα με τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου προσπαθούμε να προωθήσουμε τη συμφωνία για τις επενδύσεις. Εάν κάποτε τεθεί σε λειτουργία μια τέτοια συμφωνία είναι σαφές ότι θα μας βοηθήσει να έχουμε την απαραίτητη αμοιβαιότητα ε, στον τομέα των επενδύσεων. Και επίσης ε, και το θέμα των επιδοτήσεων Ε, που προσφέρει η Κίνα στις ε, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των ενδιαμέσων χωρών σε κάποιους από τους διαδρόμους αυτούς από όπου μεταφέρονται εμπορεύματα κινέζικα προς την Ευρώπη. Θα θέλαμε λοιπόν να ε, καταργηθούν τέτοιου είδους συμφωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας. Σε κάποιους τομείς μας πιέζουν τα κράτη-μέλη. Όλες οι χώρες μέλη νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ότι είναι σωστό να προωθήσουμε σε κάποιες μορφές συνεργασίας αλλά η συνεργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται σαν ενιαία κατά κάποιο τρόπο ε, πλευρά ιδιαίτερα όταν έχουμε τόσο μεγάλους εμπορικούς εταίρους απέναντί μας. Στα πλαίσια της πλατφόρμας για τη συνδεσιμότητα και πέρα από την Κινεζική και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής είχαμε εκπροσώπους από όλες τις χώρες μέλη Επίσης είχαμε τις ενώσεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας, εκπροσώπους της Ανατολικής Γειτονίας, είχαμε μια αντιπροσωπεία υπουργική από την Ουκρανία. Θα προσκληθούν και στην επόμενη συνάντηση της πλατφόρμας και είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν μέρος. Θέλω να πω ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα προγράμματα και σε συγκεκριμένες ευκαιρίες. Και εγώ αναφέρομαι κυρίως σωστής μεταφορές, αλλά είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν αντίστοιχες άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες και σε άλλους τομείς πρέπει όμως να έχουμε την πλήρη στήριξη των κρατών μελών. Θα πρέπει να συνεργάζονται μαζί μας και μεταξύ τους τα κράτη-μέλη και στο Πεκίνο και φυσικά εδώ, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να πετύχουμε τους στόχους. Καλώς, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να δώσει κάποια απάντηση. Ένα σχόλιο μόνο. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα εμπειρογνώμων στα θέματα του εμπορίου, αλλά στην ερώτησή σας για το αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ε, με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ίσως όχι ακόμα. Ίσως να είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο γιατί έχουμε μεταξύ μας πολλές διαφορές, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και να βρούμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε να προσδώσουμε περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή πολιτική για την Ασία. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε μια θεωρητική, αν θέλετε, σε ένα θεωρητικό επίπεδο που βασίζεται σε συγκεκριμένες κοινέ αξίες, αλλά θα πρέπει να δούμε εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που θα ευνοήσουν να βελτιωθεί η συγκεκριμένη αυτή ε, προσπάθεια. και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πόσα χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε, με πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε μέρος Μιλήσατε για την λεγόμενη εργαλειοθήκη. Εγώ μιλάω από, θα έλεγα, μιας περιορισμένης πλευράς την εικόνα που έχουμε σε σχέση με, τον, με τη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας που έχουμε στην διάθεσή μας. Τώρα, σε σχέση με την τεχνολογία η οποία είναι διαθέσιμη στην παρούσα φάση, να πω ότι στην ουσία βρισκόμαστε σε ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Για να το πετύχουμε απαιτείται μια εργαλειοθήκη η οποία να επιτρέπει σε νέες επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, να μπορέσουν να τύχουν από κοινού χρηματοδότησης από πλευράς των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να πετύχουμε αυτές τις οικονομίες κλίμακας που θέλουμε. Ε, προς το παρόν το 5G, το 5G είναι ε, ένα τεχνικό στάνταρ, αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε πάνω σε αυτό να βασίσουμε τις νέες τεχνολογίες και να χτίσουμε. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα αν θέλουμε να διατηρήσουμε ε, στην Ήπειρο την Ευρωπαϊκή τις δυνατότητες καινοτομίας και έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Κίνα με ένα ισότιμο τρόπο. Αυτά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τα μέλη του πάνελ, ευχαριστούμε και εσάς. Ένα ερωτηματικά μου δημιουργήσατε. Μερικά τα απαντήσατε είναι το θέμα αυτό της διασύνδεσης, των δυνατοτήτων διασύνδεσης. Τι μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ και όχι μόνο. Και πάλι σας ευχαριστώ και καλό ταξίδι.